τη συζήτησή μας σχετικά με την εμπορική πολιτική, θα πρέπει να σας πω μερικά πραγματάκια. Πρώτον, εγκρίνουμε την μύρηση διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι, οπότε εγκρίνεται. Έγκριση των πρακτικών των προηγούμενων συναντησών μας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Σημείο 4. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Οι συντονιστές αποφάσισαν στις 10 Οκτωβρίου για κάποια θέματα τα οποία σας ανακοινώνονται και εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνονται. Και εννοείται αυτή η συνεδρίαση ως ήθιστε αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο. Οπότε καλώς ήρθατε από τη Λισαβόνα στο Γκέτεμπορκ, από Θεσσαλονίκη και βεβαίως έχει, υπάρχει και διερμηνία. Και γι' αυτό να μιλάτε παρακαλώ καθαρά και όχι πάρα πολύ γρήγορα. Και έτσι φτάνουμε τώρα στη συζήτηση που θα έχουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ πέρα πολλούς εμπειρογνώμονες και την Επίτροπο. Είναι η τρίτη φορά που η Επιτροπή Ίντα οργανώνει μια τέτοια ακρόαση για την εμπορική πολιτική. Και είναι πραγματικά αναγκαίο ε, να καθίσουμε να συζητήσουμε και να σκεφτούμε και να προβληματιστούμε για την ε, στρατηγική που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι ότι θα συζητήσουμε αυτή η νέα στρατηγική, τι έχει προσφέρει στον κόσμο, ποια είναι τα ωφέλη για τους πολίτες μας. Εννοείται ότι και το περιβάλλον γύρω από το εμπόριο έχει αλλάξει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και μερικές φορές η στρατηγική μας πρέπει να προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα στις νέες προκλήσεις που έχει μπροστά της. Είχα σκεφτεί ότι αυτού του είδους η συζήτηση θα πρέπει να είναι πραγματικά μια συζήτηση και όχι μονόλογοι και παρουσιάσεις. Γι' αυτό και αυτή τη φορά αποφασίσαμε να οργανώσουμε τη συζήτηση κάπως διαφορετικά από ό,τι το κάναμε τις δύο προηγούμενες φορές. Και είμαι πολύ τυχερός που έχω τον Άλαν Μπίτι, ο οποίος δέχτηκε να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή σήμερα. που είναι κύριος αναλυτής στους Financial Times με έδρα της Βρυξέλλες και είναι πυρογνώμων σε θέματα εμπορίου και οικονομίας. Εκείνος λοιπόν θα αναλάβει το συντονισμό της συζήτησης, που θα είναι πολύ ζωντανή φαντάζομαι, ανάμεσα στους εμπειρογνώμονες και τους ευρωβουλευτές φυσικά, αλλά επίσης και μία ομάδα φοιτητών που έχουμε εδώ από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Μερικές φορές το εμπόριο είναι μέσα σε μία φούσκα στη φούσκα της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΙΝΤΑ. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να ακούμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια και απ' έξω. Οπότε καλώς ήρθαν εδώ οι φοιτητέ από τα δύο αυτά πανεπιστήμια. εναρκτήριο λάκισμα τώρα. Η Επίτροπος Μάλστρομ είναι μαζί μας και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καλησπέρα και σας ευχαριστώ που με καλέσατε και πάλι σε αυτή την ημερίδα που οργανώνεται για την εμπορική πολιτική. Την τελευταία φορά όταν μίλησα για το Trade for All, είπαμε ποιοι είναι οι στόχοι, τι περιμένουμε. Τότε ήμασταν μόνο στην αρχή. Τώρα βέβαια αλλάζει το πρόσωπο του εμπορίου. Τα τελευταία χρόνια είχαμε να κάνουμε πολλά στο εμπόριο είχαμε μια ημερήσια διάταξη πολύ φιλόδοξη για διαπραγματεύσεις. Από πέρυσι εφαρμόζεται η συμφωνία με τον Καναδά, έχουμε διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ, έχουμε πολιτική συμφωνία με το Μεξικό, ε, Τώρα τελειοποιούνται τα τεχνικά ζητήματα. Πήγα επίση στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία το καλοκαίρι για να αρχίσουν διαπραγματεύσει και μαζί του. Και άρχισε επίση και συνομιλίε με, για την προσχώρηση στο European Song Contest της Νέας Ζηλανδίας. Εντάξει, μπορεί να μην είναι εμπορικό ακριβώς, αλλά ναι. Επίσης έχουμε με τη Χιλή, την Ινδονησία, ε, συνομιλίες και έχουμε ξεκινήσει και μία διαπραγμάτευση για την προστασία των επενδύσεων με την Κίνα. Όλα αυτά τα έχουμε στο τραπέζι μπροστά μας λοιπόν. Θέλουμε επίσης να ενημερώσουμε κάπως και τα εργαλεία που διαθέτουμε για περιπτώσεις ελέγχου ασφάλειας σε θέματα εμπορίου. Και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από το καλοκαίρι, με τη βοήθεια, ε, το Χριστούγεννα, συγγνώμη, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, για θέματα διαφάνειας. Έχουμε ασχοληθεί πολύ και προσπαθούμε τα ωφέλη του εμπορίου να τα διευρύνουμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη στο εμπόριο που τόσο πολύ χρειάζεται. Στηρίζουμε τις αρχίες και τις αξίες μας και θέλουμε ένα περιβάλλον με ωφέλη για όλους. Δεν είναι εύκολο, αλλά το προσπαθούμε. Ποιες είναι οι προκλήσεις τώρα που έχουμε μπροστά μας. Πριν ε, παγιωθεί η εμπορική πολιτική μας ε, εδώ, πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε και τη σταθερότητα στο διεθνέ εμπόριο. Και ένα από τα πρώτα ζητήματα είναι να υποφελωθούμε όσο γίνεται περισσότερο από τις συμφωνίες. Και εδώ έρχεται το θέμα του πώς ε, τίθεται σε εφαρμογή μια συμφωνία. Γιατί το να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις χωρίς όμως να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή, στην πράξη δεν έχει νόημα. Είναι σαν να μαθαίνεις κάποιον οδήγηση χωρίς να το βάλεις στο αυτοκίνητο να οδηγήσει. Οπότε λοιπόν πρέπει να εκτιμήσουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να βελτιωθεί για να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον και να έχουμε καλύτερα επιχειρήματα για το εμπόριο. Επίσης, προβάλλουμε και περισσότερο με αυτό τον τρόπο το τι ακριβώς κάνουμε. Γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για την οικονομική ανάπτυξη και τους δασμούς, πρόκειται και για τις αξίες μας. Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ οι δικέ μας οι προδιαγραφέ να υπάρχουν σε εμπορικέ μα συμφωνίε. είτε πρόκειται για τα τρόφιμα, είτε πρόκειται για το περιβάλλον. Όλε οι συμφωνίε έχουν ε, δεσμευτικέ ρήτρε για αυτά τα θέματα. Γιατί σε αυτή τη θητεία άλλαξαν οι εμπορικέ συμφωνίε. Δεν πρόκειται μόνο για την οικονομία μα, παρόλο που είναι κάτι πολύ σημαντικό, αποτελούν και μέσο διάδοση των αξιών μα. Συνεπώ, οι εκθέσει μα, σαν και αυτέ που σα παρουσιάζουμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό και αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για τη διαφάνεια. Είμαστε ε, αυτός που διαπραγματεύεται με περισσότερη διαφάνεια από ότι οποιοδήποτε άλλο ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι ο κόσμος έγινε πιο ανοιχτός και είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Επίσης η έκθεση για την εφαρμογή των συμφωνιών γίνεται περισσότερο ανοιχτή. Έχουμε 25 συμφωνίες με 62 εταίρου. έχουμε τις παλιές συμφωνίες όπως εκείνη με το Μεξικό, τη Χιλή και τις χώρες της Μεσογείου, αλλά έχουμε και νέες όπως με την Νότια Κορέα και τον Καναδά. Έχουμε παντό είδου από τις ε, ε, συμφωνίες ε, ελεύθερου εμπορίου με τους γείτονές μας, μέχρι και τις άλλες που είναι με την Αφρική και τον Ειρηνικό. Αυτό με δύο λόγια. Τώρα θα σας πω πού έχουμε καταλήξει. Και θα αναφερθώ και πού διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και πώς θα το πετύχουμε αυτό και πώς όλα αυτά μπαίνουν στο γενικότερο πλαίσιο της εμπορικής μας στρατηγικής. Λοιπόν, πού έχουμε καταλήξει προς το παρόν. Ότι αξίζει τον κόπο το εμπόριο. Οι συμφωνίες μας εξακολουθούν να ενισχύουν ε, τις εξαγωγές μας βλέπουμε θετικές τάσεις. Με την Νότια Κορέα έχουμε αύξηση του εμπορίου πάνω από 12%, με την Κολομβία 11%, Κεντρική Αμερική γενικώ 7%. Και έτσι αντιστρέφονται οι αρνητικές τάσεις που είχαμε νωρίτερα. Από τη συμφωνία με τον Καναδά είναι νωρίς ακόμα. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως, δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα αρκετά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν θετικές τάσεις ήδη. Μηχανήματα, Εφαρμογέ, υπάρχει αύξηση 8%, φαρμακευτικά 10% και γενικά το εμπόριο έχει αυξηθεί σε κάτι παραπάνω από 7%. Οπότε οι συμφωνία ΣΕΤΑ που έχουμε με τον Καναδά κόβει 98% των δασμών για αγαθά και υπηρεσίες, μεταφορές, ταξίδια, ασφάλεια, επικοινωνία. Όλοι αυτοί οι κλάδοι εποφελούνται από τη συμφωνία ΣΕΤΑ. Τώρα, για τους εμπορικούς δασμού, Οι εμπορικές μας συμφωνίες αντιμετωπίσουν το θέμα των δασμών για προϊόντα για την υγεία με την Ουκρανία έχουμε επίσης για παλιοσίδερα επίσης με το Περού δεν έχουμε πια δασμούς για πολλά στην Καναδική Συμφωνία επίσης σταδιακά άρουμε του θεσμούς για 91% των αγροτικών μας προϊόντων εξακολουθώντας όμως να προστατεύουμε τα πιο ευαίσθητα αγροτικά μας προϊόντα. Οπότε οι εμπορικές συμφωνίες αποφέρουν καρπούς για τη Γεωργία. Από τότε που άρχισε η συμφωνία μας με την Νότια Κορέα, 10% έχουν αυξηθεί η εξαγωγή μας ε, στα αγροτικά προϊόντα. Το 1 τρίτο των προϊόντων καλύπτονται από τέτοιε συμφωνίε. Είναι κάτι καλό για τι επιχειρήσει μα, είναι κάτι καλό για του καταναλωτέ. Προστατεύουμε επίση τη γεωργία μα και τα προϊόντα μα μέσω των γεωγραφικών ενδείξεων για να δείξουμε ότι υπάρχουν κάποια τοπικά προϊόντα τα οποία πρέπει να προστατεύονται. Και το κάνουμε αυτό. Οι συμφωνίες λοιπόν προσφέρουν ευκαιρίες στη Γεωργία. Εξακολουθούμε να έχουμε υψηλέ προδιαγραφές ασφάλειας βέβαια και για το περιβάλλον. Και ακριβώ αυτά είναι τα κεφάλαια που αναφέρονται στην αηφόρα ανάπτυξη. Τώρα κοιτάμε πώ θα εφαρμοστούν όλα αυτά με ένα σχέδιο 15 σημείων που αφορά όλε τις χώρες. Εδώ συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Γιατί από εκείνη μαθαίνουμε ακριβώ ποιε είναι οι επιπτώσεις. Για το Περού και την Κολομβία βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο άνοιγμα σήμερα από ό,τι κατά το παρελθόν. Πολλά έχουν γίνει. Τώρα, το 2017 οι εξαγωγές μας θα μπορούσαν να είχαν υποφεληθεί από 3,3% παραπάνω εξοικονόμηση από τους δεσμούς. Συνεπώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα επικεντρωνόμαστε στην διάδοση των ωφελών πολύ περισσότερο και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι το 99% των επιχειρήσεών μας που προσφέρουν 85% των θέσεων απασχόλησης. Συνεπώς πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα και να περάσουν στις ξένες αγορές. Χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση, ε, βάσεις δεδομένων, υπάρχει ένα help desk για το εμπόριο και να ανοίξουν οι αγορές για τους πιο μικρούς φορείς γιατί δεν μπορούν να τα καταφέρουν με τους δασμούς. Καταλαβαίνετε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο από ό,τι μεγάλες. Τώρα, στις διαπραγματεύσεις με το Καναδά, βήμα-βήμα είχαμε κατευθύντες γραμμές για να εξηγήσουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συμφωνία μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με επιτυχία. Και θέλουμε να το συμπεριλάβουμε αυτό και σε επόμενες συμφωνίες, με την Ιαπωνία. Για παράδειγμα, ενισχύουμε και τη συνεργασία μας με τις χώρες μέλη μέσω της νέας μας ομάδας της συντονιστικής για τέτοιες εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε πληροφορίε και πραγματογνωμοσύνη. Συζητάμε την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων για τα εργασιακά και για το περιβάλλον και ανταλλάσσουμε πληροφορίε. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει με τι διάφορε κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπίες και φυσικά και ο καθένα στην εκλογική του περιφέρεια. Τέλος όλα αυτά είναι καλά. Δημερός, πολύ καλά, διευκολύνουμε το εμπόριο, αλλά η μεγάλη πρόκληση είναι να προστατεύσουμε το πολυμερές σύστημα, των ΠΟΕ. Τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθούμε στην εφαρμογή των συμφωνιών, αλλά και η αναζωγόνηση του ΠΟΕ, έτσι ώστε να έχουμε παγκόσμιους κανόνες που να λειτουργούν και να γίνονται σεβαστοί. Για δεκαετίες βοήθησε ο ΠΟΕ και άνοιξαν οι αγορές και υπήρξε ολοκλήρωση των οικονομιών. Το σύστημα αυτό όμως σήμερα απειλείται. Όταν δημιουργήθηκε ο ΠΟΕ από τον ΚΑΤ το 1995, ο κόσμος ήταν τελώς διαφορετικός. Είχαμε 16 εκατομμύρια χρήστες στο ίντερνετ. Σήμερα έχουμε 4,2 δισεκατομμύρια. Και πολλές χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Σεδική Αραβία, το Βιετνάμ δεν συμμετείχαν στον ΠΟΕ. Ούτε καν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πω Σήμερα έχουμε 62 μέλη και το 95 τα περισσότερα οικονομικά μοντέλα ήταν ίδια μεταξύ τους, ενώ σήμερα υπάρχουν διαφορετικές μορφές συμμετοχής. Κάτι που προσέφερε δυναμισμό αλλά και περιπλοκότητα, άρα πρέπει να προσαρμοστεί το σύστημα. Και μπορούμε να βοηθήσουμε. Πρώτον, πρέπει να προστατεύσουμε το σώμα επίλυσης διαφορών, γιατί αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι κανόνες δεν έχει νόημα. Δεύτερον, πρέπει να ενημερώσουμε και τον κανονισμό. Έχουμε ακόμα τους ίδιους κανόνες που είχαμε και το 95, ελάχιστα έχουν αλλάξει. Εδώ πρέπει να προχωρήσουμε. Και τρίτον, πρέπει να ενισχύσουμε την διαδικασία του ΠΟΕ, αυτή καθεαυτή, για να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και να υπάρχουν διαδικασίες που θα επιλύουν τις εντάσεις σε πρώιμο στάδιο. Συνεπώς χρειάζεται συνεργασία με όλες τις χώρες παγκοσμίω για να καταλήξουμε σε προτάσεις που θα ενημερώσουν, θα εξυγχρονίσουν και θα ενισχύσουν τον ΠΟΕ, ώστε να αποτελέσει έναν οργανισμό κατάλληλο για τον 21ο αιώνα. Σίγουρα ζούμε σε έναν κόσμο περίπλοκο, με πολλές γεωστρατηγικές αλλαγές, απειλές, αναδιόμενες δυνάμεις, περιβαλλοντικές καταστροφές, μεγάλη αβεβαιότητα Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε για να προετοιμαστούμε για όλα αυτά. Ε, μπορούμε να έχουμε οικονομική σταθερότητα στις χώρες μας, εφαρμόζοντας τις εμπορικές συμφωνίες, γιατί από αυτές ε, ξεκινάει το οικονομικό όφελος. Και πρέπει να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης και ευημερία. Να εφαρμόζουμε επίσης τα κεφάλαια που έχουν να κάνουν με την αηφόρο ανάπτυξη με τρόπο που πραγματικά να προσφέρει αηφόρο ανάπτυξη σύμφωνα με τις αξίες μας. Και στο εξωτερικό πρέπει να υπερασπιστούμε την πολυμερή τάξη. Πρέπει να στηρίξουμε την αναζωγόνηση του ΠΟΕ. Και εδώ εξαρτώμεθα από εσά, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα μεγάλο βαθμό και σας είμαστε ευγνώμονες προς το παρόν. Αλλά <clears throat> όλοι μπορείτε να βοηθήσετε. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό για να διασφαλίσουμε τη δικιά μα θέση στον κόσμο ως εμπορικό παράγων στον 21ο αιώνα. Ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπο. Το όνομα μου είναι ε, Τζον Πίτι και εργάζομαι για τους Financial Times. Γράφω για το εμπόριο εδώ και 15 χρόνια. Με κειμενόμενη συχνότητα. Και πρέπει να πω ότι κάποτε ήταν ένα θέμα πολύ διαφορετικό από ό,τι σήμερα. Μέχρι πριν από τρία χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα Trade for All, Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η γενική εικόνα ήταν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εσωτερικέ αναταράξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη. Υπήρχε πολλή ανησυχία για το τι γίνεται με το εμπόριο εσωτερικό και χρειαζόταν περισσότερη συμμετοχή όλων. Αυτό τώρα φαίνεται ότι ήταν μια χρυσή εποχή, διότι το Trade for All πρέπει να λειτουργήσει ενώ διεξάγεται και μένεται ένα παγκόσμιο πόλεμο ε, στο εμπόριο με πρωταγωνιστές στην Κίνα και την τη ΣΥΠΑ. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι κάνουμε τώρα, τι μπορεί να γίνει τώρα για το εμπόριο και πώς μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί. Εδώ έχουμε ένα πάνελ για να περάσουμε στι ενδεχόμενε απαντήσει σε αυτό το θέμα. Θα γίνουν κάποιες παρουσιάσεις, μπορούν να υπάρξουν ερωταπαντήσεις και από το κοινό και έτσι να καταλήξουμε σε κάποια πράγματα. Έχω δίπλα μου την ε, Εβίτα Σμιτ, την ε, κυρία Καρ, την Επίτροπο Μάλστρομ, τον ε, κύριο Λάγκε, τον κύριο Μπάρτελς, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, την κυρία Σάντος από την Business Europe και την κυρία Φερμπόβεν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας. Η πρώτη με ερώτηση είναι κάπως απλή. Από αυτή τη μεριά του πάνελ, ας πούμε. Τι διαφορά βλέπετε να έχει γίνει τα τελευταία τρία χρόνια. Πώς έχει διαμορφωθεί η εμπορική πολιτική και πώς έχει αλλάξει το πλαίσιο με το Trade for All. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κατά πρώτον. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, αν και πολλά τα είπε η Επίτροπος Μάστρομ βεβαίως, βλέπω ότι η έρευνα σε συγκεκριμένου τομεί, σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουν έχει προχωρήσει. Βλέπω να ενισχύεται η μέρημνα για τα κοινωνικά ζητήματα σε σχέση με το εμπόριο. Και κάποιες εκδηλώσεις με προβολή, όπως το βραβείο για τις εμπορικά δίκες και νόμιμες πόλεις πολλά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη τη εμπορική συμφωνία. Αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Ωστόσο, είναι δύσκολο να διεξαγάγει κανεί σαφή συμπεράσματα και να αποφασίσει ποιε είναι οι επιπτώσει στα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά ε, με τι χώρε εταίρου. Αυτό ίσω θα μπορούσαμε να το δούμε με περισσότερε λεπτομέρειε στη συνέχεια. Πολλέ βελτιώσει βλέπω στη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες στους ιστοτόπους και αυτό δεν συνέβαινε προηγουμένω, ήταν πολύ κακέ οι επιδόσει, αλλά οι επιδόσει παραμένουν χαμηλέ στο ότι ο κόσμο δεν λαμβάνει γνώση αυτών των πληροφοριών. Όπω είπε και η Επίτροπο Μάστρομ, έχει βελτιωθεί η διαφάνεια με στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, αλλά η σχέση μεταξύ διαφάνεια και εμπιστοσύνη είναι τελείω ε, χαλαρή και ασύντακτη για την ώρα. Πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Φαντάζομαι ότι τα θέματα της κοινή γνώμης και το πώς γίνεται αντιληπτή εμπορική πολιτική θα το δείτε και στη συνέχεια. Η συμμετοχή είναι κάτι που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Γίνονται πολύ περισσότερες συζητήσεις με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών πολλές συζητήσεις με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, που ούτω ή άλλως υπήρχε αλλά η κοινωνία των πολιτών πραγματικά έχει κάνει πρόοδο. Υπάρχει πλέον ομάδα εμπειρογνωμόνων. Δεν μπορώ να κρίνω πόσα από αυτά είναι πραγματικά σοβαρά και έχουν σοβαρό αντίκτυπο για την ίδια την εμπορική πολιτική και την ε, χάραξή τη. Σίγουρα ακόμη πολλά μπορούν να γίνουν, αλλά ως προς τα μέσα και τα εργαλεία μας υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Θέλετε να το αναπτύξω και αυτό τώρα. Καλά λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή και τη διαφάνεια, πιστεύω ότι ίσως θα χρειαζόταν να είμαστε ειλικρινέστεροι ως προς το τι περιμένουμε από τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών, ελεύθερου Μπορεί. Εάν δούμε τις κλασικές μελέτες αντικτύπου, συνήθω τα πορίσματά τους είναι πολύ θετικά και υπάρχει μια μεγάλη υπερβολή στο πώ διατυπώνονται. Διότι οι υπολογισμοί γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αισιόδοξα τα πορίσματα. Καλύτερα λοιπόν να ήμασταν κάπω εντυμότεροι και ειλικρινέστεροι και να λέμε ότι έχουμε προσδοκίε αλλά λίγο πιο μαζεμένε. Ε, ξέρω εγώ, το ΑΕΠ, το ΑΕΠ φορές ε, αντιμετωπίζεται με τρόπο υπερβολικό. Επίση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους κινδύνους, τα ρίσκα του εμπορίου, διότι αν θέλει κανείς να επεκτείνει το εμπόριο και τις εξαγωγές του. Σίγουρα θα υπάρξουν επιπτώσει. Αλλά μπορεί να θέλει να αναπτύξει το εμπόριο για να ενισχύσει τον ανταγωνισμό του. Οπότε αυτό σίγουρα θα πλήξει κάποια άλλα κομμάτια της οικονομίας, κάποιες θέσεις εργασία, κάποιοι τομείς τη οικονομίας θα αλλάξουν, θα ζημιωθούν. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τους χαμένους του εμπορίου, τους λεγόμενους loser. Ίσως έτσι θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Βέβαια ακούγεται πολύ αρνητικό αυτό το ποιοι είναι οι χαμένοι ή τιμένοι. Ο στόχος είναι να αποφύγει κανείς να χάνει, να έχει υπόλοιες. Ε, χρειάζονται όμως πολιτικές που θα συνοδεύσουν την μετάβαση προς μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περάσει αυτή τη δύσκολη μετάβαση, αυτό το μεταβατικό στάδιο δεν ήταν απλό, αλλά πολλές από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, επηρεάζονται κατά τις αποφάσεις των κατών μελών. Ξέρω εγώ, η εκπαίδευση, ε, τα θέματα της φορολογίας, ε, η αναδιανεμετική διάσταση του εμπορίου και της σχετικής οικονομίας. Όμως αυτά όλα οδηγούν στο πώς διαμορφώνεται η εμπορική πολιτική. Θα ήταν λοιπόν απαραίτητο να ενισχυθεί αυτός ο σύνδεσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει μόνο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο ότι τα εργαλεία των κρατών μελών και της Επιτροπής έχουν αρχίσει πλέον να είναι αλληλένδετα. Το αναφέρετε και εσείς με διάφορα παραδείγματα που είναι πραγματικές προκλήσεις για το πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. όταν άρχισα να προετοιμάζουμε για αυτή την ε, συνάντηση, ξαναπήγα στα αρχεία του υπολογιστή μου και είδα μια ομιλία που είχα εκφωνήσει εδώ στο σώμα σας το 2015 όταν συζητούσαμε την πολιτική trade for all. Μόνο και μόνο για να θυμηθώ τι είχα πει τότε. Τι λέγαμε εκείνο τον καιρό. Δυστυχώς η δική μου εικόνα για το πώς έχουν σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο θετική όπως τις προηγούμενες ομιλητρίες. Θα μπορούσα να σας πω ακριβώς τα ίδια που είχα πει τότε με τις ίδιες επικρίσεις που τότε είχα διατυπώσει. Ναι, υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά έχουμε χάσει κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες να κάνουμε σοβαρή βελτίωση και πρόοδο. Η Επίτροπος είπε ότι το εμπόριο δεν είναι μόνο οικονομική ανάπτυξη. Πραγματικά δεν είναι έτσι. Μάλιστα, στην Ευρώπη ε, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ την περίοδο που το εμπόριο ήταν συνώνυμο της οικονομικής ανάπτυξης. Αναφέρεται και άλλες αξίες, όπως το εργατικό δυναμικό. Όταν όμω αναφέρατε τα πλεονεκτήματα, Επιτροπέ, μιλήσατε μόνο για τι επιχειρήσει. Ξεχάσαμε τον κόσμο τη εργασία. Ξεχάσαμε τι αξίε που προστατεύουν τα εργασιακά δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Αυτά εξαλείφθηκαν από την ομιλία σα. Άρα, όταν κοιτάμε την στρατηγική trade for all, εμπόριο για όλου, Ισχύει ότι τα εμπορικά και τα, μάλλον τα κοινωνικά, τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά περιλαμβάνονται όντω αυτή τη στρατηγική. Όντω πραγματοποιούμε πραγματικά βήματα για να βελτιωθούν τα εργασιακά δικαιώματα του κόσμου, οι εργασιακέ συνθήκε. Μέσα από τι εμπορικέ μα συμφωνίε, που είναι ο στόχο των κεφαλαίων εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη, η ευκαιρία που πραγματικά χάθηκε ήταν να ενισχύσουμε τα κεφάλαια TST και να γίνουν πραγματικά κεφάλαια με δεσμευτικό χαρακτήρα. Ξέρω γιατί στην ΕΤΟΚ ε, έχω εκλεγεί τρία χρόνια ε, και επί τρία χρόνια συζητάμε με την Επίτροπο εάν τα κεφάλαια αυτά για του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι δεσμευτικά ή όχι. Εμεί λέμε ότι είναι πολύ αδύναμα. Οι μηχανισμοί που προβλέπονται δεν χρησιμοποιούνται. Δεν ενεργοποιούνται ποτέ. Για να μην πω για του σοβαρότερου μηχανισμού που θα έπρεπε να υπάρχουν για να ενισχύσουν πραγματικά όσα λέει το κάθε, από αυτά, το καθένα ένα από αυτά τα κεφάλαια. Και μάλιστα στο σύστημα GSP-SYN έχουμε κάποιους μηχανισμούς για να δείξουμε τα δόντια μας, όπως λένε. λένε. Στην πράξη είδαμε όμως τι συμβαίνει. Ο Επίτροπος ανακοίνωσε κατά της Καμπότζης, ας πούμε να γίνει έρευνα για το σύστημα GSP ε, χωρίς να γίνει τίποτα κατά της ε, εν λόγω χώρας. Δηλαδή, στι εμπορικές συμφωνίε μα τι γίνεται. Έχουμε βασικά εργαλεία για τον κόσμο του εμπορίου ε, που μπορούν να αντιμετωπίσουν το οποιοδήποτε πρόβλημα. Εδώ, γιατί για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξη δεν μπορούμε για το περιβάλλον και τα εργασιακά να έχουμε μηχανισμού που θα επιβάλλουν κάποια πράγματα. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια, Όπω είπα, τα ίδια θα σας έλεγα όπως σα είχα πει πριν από τρία χρόνια, αν έπρεπε να εκφωνήσω μια ομιλία. Αυτό που πραγματικά έλαξε σε αυτά τα τρία χρόνια είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερες συνομιλίες. Μιλάμε, μιλάμε εκτενώς και πάρα πολύ και συνεχώς για τα κεφάλαια αυτά, συντονίζουμε την κοινωνία των πολιτών. Στην πραγματικότητα όμως δεν βλέπω αλλαγές αυτές. Δεν τις βλέπω. Δεν τις βλέπω, πραγματικά. Υπογρέψαμε τη συμφωνία με την Ιαπωνία. Με το Βιετνάμ, αλλά ε, όντω το συζητάμε αυτό, την ελευθερία του συνασπίζεστε και του συνεταιρίζεστε, τις ελεύθερες ε, συλλογικέ συμβάσει και διαπραγματεύσει. Δεν το είδα εγώ αυτό στην εμπορική συμφωνία. Ξέρω ότι με τη είπα όταν συζητούσαμε το TTIP, ε, τότε ακόμα συμμετείχαν οι είχε συζητηθεί αυτό. Υπήρχε μια παράπλευρη συμφωνία επιτάπητο. Οι ΕΠΑ πεναχώρησαν βέβαια, ήρθηκαν τη συμφωνία από τι συζητήσει. Τα συζητάμε όμω πλέον αυτά. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Μπορεί ε, πίσω από τι κλειστέ πόρτε των συνομιλιών σα να τα συζητάτε. Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Και άμα εγώ δεν τα βλέπω, εγώ που εργάζομαι σε αυτόν τον τομέα, μάλλον δεν το βλέπει και κανεί άλλο. Έτσι. Οπότε αν πραγματικά μιλάμε για αυτά, καλό θα ήταν να τα προβάλλουμε κιόλα. Εάν μιλάμε. Για να δούμε πού θα γίνει διαφορά. Για την Νότια Κορέα επίσης. Επί χρόνια. Με τρει ε, επιτρόπου επιμπορίου. λέγαμε επιτέλου ενεργοποιήστε αυτόν τον αδύναμο μηχανισμό που υπάρχει μέσα στη συμφωνία. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Και ακόμα υπάρχουν σοβαρότατα εργασιακά δικαιώματα στην Νότια Κορέα. Και μια χαρά εμπορευόμαστε μαζί του. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε εμπορικέ μα συναλλαγέ. Θα μπορούσα να συνεχίσω με αυτό το μακροσκελή κατάλογο τέτοιων παραδειγμάτων. Μιλάμε. Μιλάμε πάρα πολύ. Έχουμε και άλλε δομέ για την κοινωνία των πολιτών για να πάρει μέρο. Αλλά κάποτε α πάψουμε μόνο να μιλάμε. Α γίνουν και τα πράγματα λίγο πράξη. Α του δώσουμε σάρκα και ωστά. Επίτροπε, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να θέλετε να απαντήσετε. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ το μέρο να επιχειρηματολογήσουμε, γιατί τα συζητάμε εδώ και τρία χρόνια στην πραγματικότητα. Αλλά εγώ νομίζω ότι έκαναν διαφορά, έκανε διαφορά η στατική μα. Δύσκολο να καταμετρηθεί βεβαίω. Εμπιστεύονται την εμπορική μα πολιτική άνθρωποι πριν από τρία χρόνια. Δύσκολο να μετρηθεί. Εγώ όμω δεν βλέπω ενδείξει ε, από το παράθυρό μου όπω έβλεπα πριν από τρία χρόνια καθημερινά. Ούτε διαδηλώσει. Αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, δεν μπορούν να γίνουν σε ένα δίμηνο. Όμω συστηματικά προσπαθούμε να ενισχύσουμε την διαφάνεια. Να γίνουν οι προτάσει μα στον βαθμό του δυνατού ε, δημόσιες. Ε, δημοσιεύουμε φυλάδια, ενημερώσεις, παίρνουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από κάθε χώρα, σε συνεργασία με τα κάτι μέλη, για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ε, στις ανάλογε εκλογικέ του περιφέρειες. Μιλάμε διερκώς με την κοινωνία των πολιτών. Σχεδόν κάθε κάτω μέλος μπορεί να στείλει πολίτε για διάλογο κάθε τόσο σε δημόσιε εκδηλώσει, όπου καθένα μπορεί να πάει και να ρωτήσει. Συζητούμε με τι εθνικέ βουλέ, τι τοπικέ βουλέ, τι περιφερειακέ βουλέ. Ε, ο διάλογο τη κοινωνία των πολιτών. Ε, Πολλέ φορέ, δεκάδε φορέ το χρόνο, έχουμε τη συμβουλευτική ομάδα. Κάνουμε πρόοδο. Όμω θέλει και χρόνο όλο αυτό. Δεν μπορούμε να χτίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου έτσι με τη μία. Δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να συμμετέχει. Ω προ τα εργασιακά, είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε. Και πριν υπογράψουμε τη συμφωνία με τον Καναδά, ο Καναδά είχε προσχωρήσει σε κάποιε συμφωνίε, συμβάσει του ILO, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασία, που δεν είχε σκοπό να το κάνει προηγουμένω. Τα επιτάχυνε. Και βεβαίω συζητάμε τα εργασιακά ζητήματα με το Βιετνάμ. Τα έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Αλλά υπάρχουν και περιορισμοί. Από μια εμπορική συμφωνία δεν μπορούμε να βγάλουμε καινούργια εργασιακά δικαιώματα για την κάθε χώρα. Ούτε μπορεί να αλλάξουμε το εργασιακό του δίκαιο. Ε, κάποια πράγματα μπορεί να προσαρμοστούν, όχι όλα όμω. Αναφέρατε την Καμπότζη, το είπατε και μόνοι σα. Είχαν γίνει ήδη κάποιε κινήσει στον τομέα των εργασιακών και τη ελευθερία του λόγου. Όμω, υπάρχει ο μηχανισμό GSP. Ε, πιέζουμε, πιέζουμε την Κορέα, πιέζουμε το Περού. Υπάρχουν και εκεί κάποιες κινήσεις. Κινούμεθα, θα λοιπόν, αλλά χρειάζεται χρόνος. Υπάρχει πραγματική δράση και στις χώρες αυτές ε, και είναι εταίροι. Ε, συζητούμε μαζί τους, συνομιλούμε αλλά χρειάζεται χρόνο. Και πάλι η εμπορική πολιτική δεν μπορεί να είναι το μόνο εργαλείο για να μεταμορφώσουμε τον κόσμο σε κάτι υπέροχο. Πρέπει και άλλοι να έχουν διάθεση και μπορεί να είμαστε ρεαλιστέ ότι μπορεί να πετύχουμε μια εμπορική συμφωνία. Έχουμε και την πολιτική την εξωτερική. Έχουμε την πολιτική συνεργασία στην και βοήθεια. Όλα αυτά είναι μέρο τη ίδια διαδικασία. Όμω εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά τα τελευταία 7 χρόνια. Και είναι λίγα τρία χρόνια, έτσι. Δεν είναι πολύ καιρό. Πιέζουμε. Πιέζουμε για να προχωρήσουν όλα αυτά. Εγώ βλέπω κάποια αποτελέσματα. Ε, θέλουμε κι άλλα, δεν λέω. Αλλά είναι καθημερινή η δουλειά μα και έχουμε περιβαλλοντικέ συμφωνίε, μνήε στη Συμφωνία των Παρισίων σε όλε μα τι εμπορικέ συμφωνίε, την αρχή τη προφύλαξη που αναφέρεται αναφέρεται στι εμπορικέ μα εφορίε αυτέ. Αλλά πρέπει και άλλε χώρε να κοιτάξουν να τα υλοποιήσουν όλα αυτά. Όμω διαδίδουμε αυτέ τι αξίε. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προοδευτικοί, διορατικοί, βιώσιμοι. Δεν ξέρω πώ να την εμπορική μα πολιτική. Πρέπει και άλλε χώρε να θέλουν τα μέτρα αυτά στι εμπορικέ του δράσει. Yeah, or... Ναι, είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι. Σίγουρος δεν είμαι. Βεβαίω το σίγουρο είναι υπήρξαν αλλαγές το τελευταίο διάστημα. Ε, όταν εγώ ανέλαβα τα καθήκοντα του Προέδρου, μόνο 23, ε, 23 ευρωβουλευτές είχαν πρόσβαση στα έγγραφα της διαπραγμάτευσης. Τώρα πλέον η πρόσβαση αυτή είναι γενική και έχουμε πλέον συμφωνία ότι η διαπραγματευτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύεται πλέον στην ισοσελίδα κτλ. κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αλλαγές ε, ως προς τη διαφάνεια αλλά και ως προς τις θέσεις. Θυμάμαι ότι ε, στο παρελθόν η Κομισιόν επέμενε στο τοξικό σύστημα του ISDS, το οποίο πλέον έχει εγκαταλειφθεί, προκρίνονται τα δικαστήρια. Σημειώνεται πρόοδος λοιπόν. Από την άλλη πλευρά βεβαίως ε, συνεχίζεται ο διάλογος για το κεφάλαιο TST, για την στενότερη συνεργασία με άλλους τομείς πολιτικής. Υπάρχουν σε κάθε περίπτωση περιθώρια βελτίωσης. Βελτίωσης που είναι απαραίτητη, γιατί το διεθνές εμπορικό περιβάλλον έχει αλλάξει θεμελιωδώς. Πριν από τρία χρόνια δεν θα πω ότι τα πάντα ήταν μια χαρά, αλλά μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η επικέντρωση λοιπόν σε ένα δίκαιο σύστημα για το εμπόριο που θα βασίζεται σε κανόνες και θα εξασφαλίζει πρότυπα θα σέβεται προδιαγραφές, θα εξασφαλίζει χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές, είναι πραγματικά μια νέα διάσταση της συνολικής συζήτησης που γίνεται. Και τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι το εξή. Μπορούμε να συνάψουμε εμπορικές συμφωνίες, να χαράσουμε εμπορικο, εμπορική πολιτική εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κάποιες φορές οι προσδοκίες για αυτές τις συμφωνίες είναι πολύ υψηλές. Κάποιοι περιμένουν ότι θα λύσουν ακόμη και προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λύσουν εμπορικές συμφωνίες. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας και να εξασφαλίσουμε κατά συνέπεια μεγαλύτερη συνοχή με άλλες πολιτικές μας, σε άλλους τομείς πολιτικής ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Κατά τη γνώμη μου, σε κάθε περίπτωση το ποτήρι είναι μισογεμάτο. I mean, difficult to know how to είναι δύσκολο να μετρήσει κανείς την, ε, τις βελτιώσεις που έχουν υπάρξει ή την πρόοδο, όπως είπαν και προηγούμενοι ομιλητές. Και είναι δύσκολο να μπορεί κανείς να ε, προβλέψει ε, ποιες και τι είδους θα είναι οι αλλαγές που θα προκύψουν. Βεβαίως, από το εμπόριο υπάρχουν, στο εμπόριο υπάρχουν πάντοτε κερδισμένοι και χαμένοι. Η ε, γραφειοκρατία βεβαίως είναι αυτή που ωφελείται ε, εκτός αν ε, ε, συμφωνήσουμε ότι το εμπόριο πραγματικά είναι ένα στοιχείο της, που έχει στα χέρια της η παγκοσμιοποίηση και που αναγκαστικά οδηγεί κάποιους εκτός αγοράς εργασίας. Πρέπει κανείς να, να, να αναδιατυπώσει λοιπόν το trade for all. Για μένα το trade for all σημαίνει εμπόριο για όλους τους Ευρωπαίους, όχι εμπόριο για όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι από την Αυστραλία, ζω στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζω ακόμη δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οπτική μου είναι ίσως λίγο διαφορετική. Ποια ήταν η διαφορά που επέφερε αυτό το πακέτο του εμπορίου για όλους. Μπορώ να σας πω το εξή. Συνέβαλε σημαντικά στο άνοιγμα μιας συζήτησης στον κόσμο για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης και αυτό δεν είναι καινούριο. Ε, και η ίδια ίδρυση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας γύρω από αυτό το ζήτημα ε, κινούνταν. Όμω, η στρατηγική που έχει υιοθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρόμοια με εκείνη που έχουν υιοθετήσει άλλε χώρες. Συγκεκριμένα, να επιβάλλεις τα δικά σου ρυθμιστικά πρότυπα σε άλλες χώρες, στους εμπορικούς σου εταίρους. Και αυτό είναι δύσκολο διότι μπορεί να έχεις εσύ ε, ε, κανονιστικά πρότυπα τα οποία μπορεί να μην τα θέλουν να τα δεχτούν οι εμπορικοί σου εταίροι. Γι' αυτό και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε μακροπρόθεσμα να ε, παρακινήσει και άλλες χώρες να εντάσσουν όρους και κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη που αντανακλούν κυρίως ε, τις επιθυμίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες φορές επικοινωνούν και με ορισμένα διεθνή πρότυπα, αλλά όχι πάντοτε. Και κάποιες φορές γίνεται και με, με κρυφούς τρόπους, όχι μόνο με, την, με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από μια, ε, από μια σύμβαση. Πολλέ φορές ε, αυτά ε, εμφανίζονται μέσω της εταιρική κοινωνικής ευθύνη των ετικετών οικολογικής ε, προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τη γνώμη μου, Το να υπάρχει μια ρήτρα σε συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που θα λέει ότι το δίκαιο εμπόριο είναι αυτό που προωθείται, στην πραγματικότητα ε, προκρίνεται απλά ο ένας τρόπος παραγωγής και στην ουσία δηλαδή προστατεύεται και ένας συγκεκριμένος τρόπος παραγωγής. Άρα πρέπει κανείς να εξετάσει το σύνολο των διατάξεων αυτών των συμφωνιών για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματά τους. Και βεβαίω υπάρχει μια πολυμέτωπη, αν θέλετε, πολιτική από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και από πολλέ απόψει ήταν και επιτυχημένη συνέδεσε τα ωφέλη του εμπορίου με εκείνους που ενδεχομένως πλήττονται από τις εμπορικές δραστηριότητε. Από την άποψη ότι πολλές χώρες, άλλες χώρες, ευθυγραμμίστηκαν με τα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν φυσικά θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελειώνω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να κάνω όμως μια τελική παρατήρηση. Ότι η στρατηγική εμπόριο για όλους κατά πάσα πιθανότητα ε, είχε και ένα πολύ συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το Brexit. Ήταν και αυτό ένα από τα αποτελέσματα της, της στρατηγικής αυτής εμπόριο για όλα. Βεβαίως περιλαμβάνονται στη στρατηγική αυτή και το εμπόριο, η απασχόληση, το περιβάλλον, αλλά αποτέλεσμα ήταν και το Brexit. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Και αυτό είναι και το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο για το πώς οι εμπορικές συμφωνίες μπορεί να συνάπτονται και να εφαρμόζονται, αλλά και για το πώς εν τέλει επηρεάζουν τα πρότυπα εξαγωγών, τα συμπεφωνηθέντα βεβαίως, για το πώς πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο που μπορεί κανείς να πει στους εμπορικούς του ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά εμεί θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε τα εμπορεύματά σας από το να εισαχθούν στις, ε, στην, επικράμια, ε, στην επικράτειά μας, με όποιον πρόσφορο τρόπο βρούμε. Αυτά όλα μπορώ να πω ότι είναι ε, ίσως και μια επιτυχία του Trade for All που αποτέλεσε και μια μεταστροφή ε, ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζει το, ε, το εμπόριο. Ως Βρετανός ε, μετράω τις φορές που αναφέρεται το Brexit, το Brexit την, την ώρα που περνά μέχρι κάποιος να αναφέρει το Brexit. 47,5 λεπτά μας πήρε σήμερα. Ε, ευχαριστώ. Τι Λουίς Σάντος. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που αναφέρθηκαν πριν για τις αλλαγές που έχουν προκύψει. Η μεγαλύτερη ίσως όχι εξαιτία του Trade for All, αλλά εξαιτία του περιβάλλοντος είναι ότι το εμπόριο έχει γίνει το πρώτο θέμα στην παγκόσμια ημερήσια διάταξη. Πριν ήταν ένα τεχνικό ζήτημα, τώρα είναι γκάρσιο. Αυτό είναι ένα. Και είναι καλό, γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται περισσότερο το εμπόριο, όλοι το συζητούν, ακόμα και οι άνθρωποι, οι απλοί που παλιά δεν συζητούσαν και δεν έχουν σπουδάσει για το εμπόριο, το συζητούν. Έπειτα υπάρχει και πίεση, γιατί η ζήτηση για εμπόριο είναι μεγαλύτερη. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχει αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα αλλά έχει γίνει και αντικείμενο παζαρέματος, που και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Όταν συζητάμε για κυρώσεις σήμερα, συζητάμε για κάτι που έχει επιπτώσει στο εμπόριο. Συνεπώς όλο και περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν το εμπόριο ως πολιτικό εργαλείο. Τώρα το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας είναι το εξής. Αυτό βοηθάει Μπορώ να συζητήσω με τη Λίνα κατά πόσο επηρεάζει εξίσου επιχειρήσεις, τα εργαζόμενους, ε, της ή πολιτών. Πρώτα απ' όλα, προσφέρει στις επιχειρήσεις. Προσφέρει με την έννοια ότι έχουμε περισσότερες εμπορικές συμφωνίες, πολλές από αυτές έχουν κυρωθεί και μένει τώρα να τεθούν σε εφαρμογή Οπότε το βάρος πέφτει ακριβώς στην εφαρμογή, στην πράξη, γιατί η Κομισιόν διαπραγματεύεται. Τώρα εμείς πρέπει να φροντίσουμε για την υλοποίηση. Το Trade for All λέμε ότι θα επιφέρει αλλαγές στο μέλλον και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε περισσότερο την ελοποίηση. Ναι, αλλά αλλάζει και ο τρόπος που πρέπει να διαπραγματευόμαστε, γιατί όταν διαπραγματευόμαστε για τους κανόνες προέλευσης των προϊόντων. Είναι ένα παράδειγμα. Ο τρόπος με τον οποίο επαληθεύονται οι κανόνες, ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να υποφεληθεί από τις προτιμήσεις, να φροντίσουμε να μην δημιουργήσουμε μια γενική συμφωνία η οποία όμως να μην μπορεί να χρησιμεύσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα η ποσότητα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κερδίζουμε και σε ποιότητα. Προς το παρόν καλά είναι τα νούμερα, αλλά τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στην βελτίωση της ε, χρήσης τέτοιων συμφωνιών, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το άλλο που θέλω να υπογραμμίσω, και είναι κάτι που υπόθηκε και πριν, ότι το εμπόριο μπορεί να προσφέρει ωφέλη απευθείας, αλλά μπορεί να έχει και κάποιες αρνητικές πτυχές, εντάξει. Αλλά το ζήτημα είναι τι θα τα κάνουμε όλα αυτά τα ωφέλη. Θα μοιραστούν εξίσου προς όλους ή όχι. Και αυτό έχει να κάνει με πολιτικές στις οποίες αναφερθήκατε κι εσείς. Δηλαδή πρέπει να έχουμε έναν συνδυασμό εμπορίου, αλλά πρέπει να έχουμε και πολιτικές. Γιατί την περιφερειακή πολιτική, τη συνοχή, ε, τα θέματα φορολογίας δεν θα τα λύσει το εμπόριο. Δεν είναι η εμπορική πολιτική που θα λύσει αυτά τα ζητήματα. Αν περιμένουμε λοιπόν από την εμπορική πολιτική να τα λύσει, τότε κοροδευόμαστε. Και στο τέλος όλοι θα απογοητευτούμε, γιατί δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Συνεπώς πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στο τι μπορεί να πετύχει το εμπόριο αλλά σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διότι θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ωφέλη από το εμπόριο και το θέλουμε το εμπόριο, το Trade for All τι προσφέρει. Μιλάμε για free trade, fair trade, δηλαδή ελεύθερο εμπόριο, αλλά μιλάμε και για το θεμητό, το δίκαιο εμπόριο. Άρα μιλάμε και για τις πρακτικές του εμπορίου. Δεν μιλάμε μόνο για το άνοιγμα των αγορών, μιλάμε και για το πώς ανοίγουμε τις αγορές. Και δεν πρόκειται εδώ πέρα μόνο για το θέμα του πόσο βιώσιμη είναι η πολιτική μας, αλλά το εμπόριο μπορεί να διορθώσει κάποια προβλήματα στην αγορά. Παλιότερα Κανείς δεν αφισβητούσε το κατά πόσο θα πρέπει να δώσουμε στην Κίνα το καθεστώς της οικονομίας της αγοράς. Άλλαξε όμως και η Κίνα, άλλαξε όμως και ο τρόπος ε, με τον οποίο εμεί αντιλαμβανόμαστε το εμπόριο. Υπάρχει αλλαγή στο περιβάλλον μας. Το περιβάλλον μας. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πάντα δικαιοσύνη για τις δικές μας επιχειρήσεις, για τους δικούς μας καταναλωτές, ότι μερικές φορές δεν ε, είμαστε όλοι στον ανταγωνισμό επίσης όρης. Και αυτά είναι θέματα που αρχίζουμε να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να το κάνουμε πολύ περισσότερο και στο μέλλον. Η κύριε Φερμπόβεν, ευχαριστώ. Εγώ μιλάω εκ μέρους της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η ερώτησή σας είναι τι διαφορές έχουν προκύψει βάσει της στρατηγικής ε, Trade for All Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής τα τρία τελευταία χρόνια. Από πλευράς του ILO λοιπόν, εμείς βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τα εργασιακά στις εμπορικές συμφωνίες ε, αυτά που τονίζουν είναι πολύ θετικά γιατί προωθούνται οι προδιαγραφές του οργανισμού μας κάτι το οποίο αποτελεί και βασικό στοιχείο του καταστατικού του ILO. Ας πούμε, κατά πολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας, της παιδικής εργασίας, πολέμηση των ε, διαφορών μεταξύ των φύλων, ε, επίσης να υπάρχει το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε κλπ. Τώρα, Παγκοσμίω βλέπουμε ότι οι προδιαγραφές εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι συμπεριλαμβάνονται σε όλες ή τόσο σε πάρα πολλές διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Το 80% ακολουθούν αυτά τα πρότυπα. Η παγκόσμια διάσκεψη για την εργασία είναι ένα τριμερές όργανο με συνδικάτα εργαζόμενους και ε, εργοδότες και κυβερνήσεις που συμφωνούν πάνω σε συγκεκριμένα πρότυπα για να υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού. Τώρα είναι αλήθεια ότι άπαξ και ως χώρα έχει κυρώσει μια συμφωνία, μετά εμφανίζονται εμπόδια. Δεν υπάρχει δηλαδή η ήπια συμμόρφωση. Και υπάρχει ένα σύστημα εποπτείας στον ILO και ένα ανεξάρτητο όργανο και του τριμερούς, της τριμερούς σύνθεσης που φροντίζει για τη συμμόρφωση στις εργασιακές προδιαγραφές. Αυτό λοιπόν που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι οι εμπορικοί εταίροι μέσω αυτού του εμπορικού εργαλείου που αναφέρει τις εργασιακές προδιαγραφές συζητούν τη συμμόρφωση και βλέπουν πού θέλουν να βελτιωθεί η εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών. Και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις που το σύστημα εποπτείας μας συνεχίζει το διάλογο με κάποια χώρα η οποία δυσκολεύει ε, την ε, εφαρμογή των προδιαγραφών μας. Οι συμφωνίες αυτές έχουν κάνει τη διαφορά και θα σας πω ένα παράδειγμα. Και μετά μπορούμε να συζητήσουμε κι άλλα, μα θέλετε. Ουσπεκιστάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Υπήρχε πρόβλημα με την εποχιακή εργασία των παιδιών στις ε, βαμβακοκαλλιέργειες. Από το 2011 μέχρι το 2015-16, πρόσφατα δηλαδή. Είδαμε όμως ότι σε δύο χρόνια περίπου με τις προσπάθειες που έγιναν και χωρίς να προθείτε το πρωτόκολλο για το βομβάκι που είναι παράρτημα στην εμπορική συμφωνία υπήρξε πίεση στη χώρα. Ο συνδυασμός τώρα αυτής της πίεσης με τις παρεμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, γιατί πήγαμε εκεί και το Μπεκιστάν αναγκάστηκε να τους συναντήσει και ήταν ευπρόσδεκτη, πριν δεν μπορούσαμε καν να πάμε. Τώρα πήγαμε. Σε λίγα χρόνια λοιπόν υπήρξε πρόοδος και η εποχιακή αυτή εργασία των παιδιών αυτές τις έξι εβδομάδες που είναι το καλοκαίρι η εργασία της βαβακαλλιέργειας, σταμάτησε. Το 2016 το Ουσμπεκιστάν είναι μια από τις τελευταίες χώρες στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή που κύρωσε όλες τις προδιαγραφές εργασίας. Δημιουργήθηκε δηλαδή συνειδητοποίηση. Και αυτό είναι κάτι θετικό. Βέβαια η διαδικασία είναι μακρά και το εμπορικό εργαλείο δεν είναι παρά ένα εργαλείο. Χρειάζονται και άλλα για να επιτευθούν καλά αποτελέσματα. Πρέπει να γίνει με τερικές σχέσεις, με συνεχή διάλογο και στήριξη. Και αυτό ακριβώς είναι στο οποίο προσβλέπει και ο Παγκόσμιος Οργασμός Εργασίας. Ωραία και για λίγα λεπτά τώρα να ακούσουμε ερωτήσεις από τους βουλευτές, επερωτήσεις θα ήθελα να θέσω την ίδια ερώτηση που έθεσε προηγουμένω στον Πρόεδρο τη Επιτροπή σα. Ε, πριν από λίγε εβδομάδε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ο κ. Τραμπ δηλαδή, άρχισαν να συζητούν το τι θα γίνει με τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους δασμούς. Ο κύριος Λάγκε, μεταξύ άλλων, είπε ότι η συμφωνία με χώρα που δεν έχει συνάψει και δεν έχει συναυθεί το όσα προβλέπουν η Συμφωνία των Παρισίων θα ήταν παράβαση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το δεδομένο, ποια είναι η περίπτωση όλα αυτά να ε, μην ε, ισχύσουν και να ξεχαστούν και να βρουν και να ξεφύγουν ε, εάν ε, υπάρξει παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Κοιτάξτε, ε, η Συμφωνία των Παρισίων είναι ε, δεσμευτική για κάθε εμπορική συμφωνία, αλλά δεν έχουμε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τι ΗΠΑ, μόνο για τα βιομηχανικά αγαθά. Οπότε δεν έχουμε συνολική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Για το λόγο λοιπόν που το αναφέρατε, είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Είπαμε με τι ΗΠΑ ότι θέλουμε ένα θετικό κατάλογο προτεραιοτήτων, αν και υπάρχουν σε πολλά πράγματα διαφωνίε. Θέλουμε όμω να επικεντρωθούμε στα θετικά. Και αυτή τη στιγμή συζητάμε κάποια ρυθμιστική συνεργασία που θα ήταν καλή για την βιομηχανία μα και την δική μα. Και βεβαίω προσπαθούμε να αποκλιμακώσουμε την ένταση που υπάρχει, να αποφύγουμε την ε, πρόβλεψη μελλοντικών δασμών και να δούμε το τι είναι, το, τι είναι τα επικοδομητικά στοιχεία που μπορούμε να ε, συζητήσουμε μαζί του. Δεν θέλουμε όμω συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Για την συμφωνία των Παρισιών δεν νομίζω θα πρέπει να εντολή για καμία μελλοντική συμφωνία χωρί ρήτρα για τη συμφωνία των Παρισιών. Ούτε θα τη ζητούσα κιόλα, έτσι. Indeed, uh, nobody knows exactly what the next... Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το επόμενο σενάριο που θα προκύψει από τη ΣΥΠΑ. Ίσως το νόημα της όλης προσπάθειας είναι κάπως να καλμάρουμε τα νεύρα όλων. Αν και δεν είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε καμιά αξιόπιστη συμφωνία με αυτήν την κυβέρνηση που τώρα κυβερνά τη χώρα. Για μένα είναι σαφές ότι θέλουν να ξαναπάρουν πίσω στις ΗΠΑ την παραγωγή. Να αλλάξει λίγο η αλυσίδα παραγωγής οξιών. και ο άλλος μεγάλος παγκόσμιος εταίρος τους θέλουν να μείνει λίγο σε χαμηλότερο επίπεδο, την Κίνα δηλαδή εννοώ. Θέλουν να προσπαθούν τα δικά τους συμφέροντα. Η μόνη δυνατότητα μιας συμφωνίας, εμπορικής συμφωνίας που να ξεκινά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε όλη αυτή την ωραία συζήτηση για το τι μέσα για το ψήφισμα. Αυτή τη στιγμή τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει εμπειρητά με τη ΣΥΠΑ συνομιλίες βεβαίως είναι προτιμότερες από τσακωμούς και εμπορικούς πολέμους. Ευχαριστώ. Ένα από τα θέματα που μπορεί να μας απασχολήσουν, πιστεύω, άκουσα πολλούς να λένε ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες από τις εμπορικές συμφωνίες. Οι εμπορικές συμφωνίες που έχουμε όμως τώρα δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε καν στην αρχική τους ε, σύνταξη ως προς την υλοποίηση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι το εμπόριο δεν μπορεί να έχει αντίκτυπο και στα υπόλοιπα ή ότι ο τρόπος που σχεδιάζονται οι εμπορικές μας συμφωνίες πρέπει να αλλάξει. Πολλά από αυτά που είπατε για τις συμφωνίες ε, οικονομικής εταιρικής σχέσης ή για το ελεύθερο εμπόριο. Δεν καλύπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά και το καθεξής. Πιστεύετε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ ή είναι πραγματικά πολύ υψηλέ προσδοκίε μας. Η μεταρρύθμιση και η αλλαγή στι εμπορικέ συμφωνίε είναι κάτι το απαραίτητο. Απ' την άλλη, όμω, όχι. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε κιόλα ή πάρα πολλά από τι συμφωνίε αυτέ. Α πούμε, αυτό που έγινε στην Καραϊβική. Εγώ πήγα 8 χρόνια ξανά και ξανά εκεί και δεν ήταν φοβερή η ε, επιρροή στην αλλαγή τη πολιτική και δεν ήταν το πρόβλημα η εμπορική συμφωνία. Βεβαίω, ε, με τι πιο δύναμε χώρε ε, ήταν τελείω ασυμμετρικέ οι συμφωνίε. Που λαμβάνουν υπόψη τι αδυναμίε των χώρων αυτών, είχε σχέση και με τη Γαλλία που χρησιμοποιήθηκαν, το πώ μπορεί να συμπεριφέρονται οι επενδυτέ ε, ω προ τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα. Προβλέπονται λοιπόν κάποιε υποχρεώσει για του επενδυτέ. Είναι μια συμφωνία με πολλέ θετικέ προθέσει. Όμω στην πράξη τελικά δεν έγιναν πολλά. Και αυτό κυρίω λόγω τη ίδια τη κατάσταση στη χώρα. Ε, και αυτό νομίζω συμβαίνει πολύ συχνά στι αναπτυσσόμενε. Οι δυνατότητε δεν υπάρχουν. Δεν μπορούν έτσι να αρπάξουν τι ευκαιρίε για να αυξήσουν τι εξαγωγέ του βάσει των εμπορικών συμφωνιών. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το δούμε. Ω προ τα εργαλεία, νομίζω μπορούμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Όπω είπα προηγουμένω, αυτό που πρέπει ακόμη να γίνει είναι να εξετάσουμε προσεκτικότερα πώς μπορούμε να αποζημιώσουμε τους loser, τους χαμένους, τους ιτημένους. Αυτό γίνεται και με τις ε, εξάντε μελέτες σκοπιμότητας και αντικτύπου. Πολλές φορές δεν είναι καλής ποιότητας, οπότε δεν χρησιμεύουν και πολύ, αλλά δεν υπάρχει και πολιτική βούληση να γίνει κάτι. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει. Όταν αυτά τα εργαλεία γίνουν καλά, αξιόπιστα, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κάτι μέλη θα πρέπει αυτό να το συζητήσουν και να εξαγάγουν τα σχετικά συμπεράσματα. Αυτό δεν συμβαίνει προ στιγμή. Κάτι άλλο σημαντικό που αναφέρεται στη στρατηγική Trade for All για την ώρα δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στο αρχικό μοντέλο, είναι η παρακολούθηση των ε, συμφωνίων ελεύθερου εμπορίου. Από αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται. Πρέπει κανεί να παρακολουθεί τι κάνουν όχι απλώ μόνο πόσε εξαγωγέ ε, και εισαγωγέ υπάρχουν και πώ αυξήθηκαν, είναι ενδιαφέρον να μελετήσει κανεί το βαθμό εμπιστοσύνη. Αλλά και τι βαθύτερε αλλαγέ που προκαλούν, πω αλλάζουν οι βιομηχανικοί κλάδοι και τομεί και η παραγωγή. Η ιδέα για την παρακολούθηση υπάρχει. Η ιδέα για τα μέσα παρακολούθησης επίση αναφέρεται. Για την ώρα όμω δεν έχει γίνει κάτι στην πράξη. Και ω προ τα κεφάλαια TST, για του στόχου τη της νομίζω ότι πολλή ενέργεια εξοδεύεται για να συνταχθούν τα κεφάλαια αυτά. Πολλέ συζητήσει, όπως είπε και η γειτονά μου. Αλλά ω προ τα αποτελέσματα έχουμε μερικά αλλά δεν αλλάζουν και τον κόσμο. Είναι λοιπόν απαραίτητο κάπως να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε και πόση προσπάθεια απαιτείται. Είναι κάποια πράγματα που μπορούμε να τα επιτύχουμε με μικρότερη προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την εξάντε ερεσιμότητα. Ζητά από του εταίρου, πούμε, να βελτιώσουν το εργατικό τους δίκαιο ή να κυρώσουν τις βασικές συμβάσει του ΕΛΟ και τα σχετικά εργασιακά πρότυπα πριν ξεκινήσει να ισχύει η συμφωνία. Οι Αμερικανοί το κάνουν, οι Καναδοί το κάνουν το ίδιο. Αλλά εφόσον η συμφωνία δεν ισχύει, ε, γιατί να υπάρχει τόση πολύ πολιτική βούληση από την άλλη πλευρά να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Κάποιες φορές ε, θέμα είναι και η έλλειψη δυνατοτήτων στις ε, χώρες εταίρους. Ε, κάτι που θα μπορούσε να υποστηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Aid for Trade, βοήθεια για το εμπόριο, να υποστηρίξει χώρε, πραγματικά να βελτιώσουν του νόμου του, πραγματικά να κάνουν αλλαγέ στην νομοθεσία του εγκαίρω και στο πώ αυτή υλοποιείται. Πέραν όμω αυτού, είναι δύσκολη η απόφαση. θέλει να ενισχύσει τι ρήτρε για τα εργασιακά Ευρωπαϊκή Ένωση στι εμπορικέ τη συμφωνίε. Διότι θα πρέπει να ε, ενισχυθούν τα κεφάλαια αυτά, αλλά να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι κι εμεί. Όταν κοιτάζα τη συμφωνία, το σχέδιο συμφωνία με την Κολομβία, πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, εκεί είπα ζητούν από την Κολομβία ε, να υλοποιήσει ένα διεξοδικότατο πρόγραμμα δράση. Έχει ένα σχετικό κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη δική τη ε, συμφωνία για τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τη δημιουργία του οικίου συμβουλευτικού σώματος. Όμω δεν πήγε πουθενά όλο αυτό. Οι Κολομβιανοί δεν ήξεραν τι πρέπει ακριβώ να εφαρμόσουν. Υπήρχε ήδη κάτι που του είχε ζητηθεί από τη ΣΥΠΑ. Εάν ζητάμε τώρα από έναν εταίρο να δημιουργήσει και άλλε θέσει εργασία για επιθεωρητέ εργασία και άλλου νόμους στο επίπεδο των φορέων που ασχολούνται με την εργασία να αυξήσει το δυναμικό και είναι αυτό προπόθεση για να συναυθεί η συμφωνία, θα πρέπει κάποιο να πάει να επαληθεύσει και να εξακριβώσει να γίνανε όλα αυτά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια απόφαση που πρέπει να τη λάβουμε. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτά. Διότι αλλάζει το τι συμφωνία έχουμε τότε και αλλάζει πολύ από το να ε, εκφράζουμε απλώ απαιτήσει επί χάρτου. Εάν θέλουμε να γίνει κάτι στην πράξη, πρέπει να υπάρξει επαλήθευση, έλεγχο, να πάνε εκπρόσωποι να συζητήσουν με την κυβέρνηση και ούτω καθεξή. Και υπάρχουν και άλλα παρελκόμενα προβλήματα που δεν θέλω καν να τα αφήξω αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο που θα μπορούσε εύκολα να γίνει ω μέρο τη εξάντια ρεσιμότητα είναι η δημιουργία ενό μηχανισμού επίλυση διαφορών για να μπορούν να αποβληθούν προσφυγέ στι χώρε που συνεργάζονται με τον ΩΣΑ ή είναι απλώ μέλη του ΩΣΑ, είναι κάτι που θα πρέπει να προβλέπετε προβλέπεται ορισμού. Διότι οι κατευθυντήριε γραμμέ του ΩΣΑ για τι πολυεθνικέ εταιρείε ζητούν την θέσπιση και τη δημιουργία των εθνικών σημείων επαφή, όπω τα ονομάζουν. Ένα μηχανισμό υποβολή προσφυγών είναι αυτό, όπου μπορεί να πάει ο πολίτη, οποιοδήποτε από την κοινότητα των πολιτών, και να πει εσεί, τάδε εταιρεία, δεν εργάζεστε, δεν ακολουθείτε τι κατευθυντήριε γραμμέ του ΩΣΕΑ και αυτό πρέπει να το δούμε. Εγώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα και εύκολα να ζητηθεί και να εφαρμοστεί. Το θέμα των κυρώσεων. Βεβαίω αυτό έχει να κάνει με το κατά πόσον υπάρχει απόφαση να συμπεριληφθεί ένα κεφάλαιο για τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά στι εμπορικέ μα συμφωνίε. Και δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι οι κυρώσει ω προ το εμπόριο επηρεάζουν αρνητικά ιδίω στο χώρο τη εργασία, τον κόσμο τη εργασία. Του εργαζομένου δηλαδή γι' αυτό και δεν φέρνουν θετικά αποτελέσματα. Οι οικονομικέ κυρώσει είναι μια ιδέα. Αλλά όχι οικονομικέ κυρώσει όπου θα πρέπει να πληρώνει ένα ποσό η χώρα, συμβαλόμενη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώ εάν η χώρα εταίρο δεν ακολουθεί τις αρχές των εργασιακών όπως προκύπτουν από την εμπορική συμφωνία και δεν τις υλοποιεί ακολούθως, θα πρέπει να, υποβάλει, να πληρώνει κάποια πρόστιμο. Και αυτό το πρόστιμο να πηγαίνει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στον κόσμο της εργασίας και στους εργαζομένους στην εν λόγω χώρα. Και κάτι τελευταίο, διότι με ρωτήσατε τι γίνεται με τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω σημαντικό είναι αυτό να το δούμε και από μια ευρύτερη οπτική γωνία. Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει μια εμπορική συμφωνία, σίγουρα. Και υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη που πάνε πέρα από τι εμπορικέ συμφωνίε, όπω η φοροδιαφυγή, οι κλιματικέ αλλαγέ. Η Αφρική χάνει πάρα πολλά λόγω τη φοροδιαφυγή. Οι επιδοτήσει, η παραοικονομία και άλλοι τομεί. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Εν μέρη, επηρεάζουν περισσότερο από ότι τα ίδια τα εμπορικά ζητήματα. Ωραία. Θα σα ξαναδώσω το λόγο σε λεπτά. Απλώ να το θέσω και στη Λουίζα τώρα το ίδιο. Λουίζα, όταν ακούτε όλε αυτέ τι φοβερέ ιδέε για την εξάντερη αιρεσιμότητα και για όλο και περισσότερε προποθέσει και όλο και περισσότερα κεφάλαια που περιλαμβάνονται στι εμπορικέ συμφωνίε, μόνοι σα είπατε ότι περιμένουμε πάρα πολλά από αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε. Πιστεύετε ότι έχουμε βάσει τον πύχη πολύ ψηλά και ότι επιβαρύνουμε τι εταιρείε και τι επιχειρήσει με πρότυπα και προδιαγραφέ που δεν θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν τους ε, επιδιωκόμενους στόχους. Απλώς θα τους ε, φορτώσουν περισσότερο φόρτο εργασίας. Όπως ε, είπα, εμείς θέλουμε και την ποσότητα, αλλά θέλουμε και την ποιότητα. Κατά την έννοια ότι δεν αρκεί να αυξάνονται οι εξαγωγές μας. Είναι εξίσου σημαντικό να ωφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις από την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών. Και βεβαίως ε, οι διαπραγματεύσεις γύρω από τις συμφωνίες αυτές είναι πάρα πολύ περίπλοκες. Γιατί βεβαίως δεν είμαστε μόνοι μα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Βεβαίως καλό είναι να υπάρχει ένα πρότυπο όσον αφορά αυτές τι εμπορικέ συμφωνίε, αλλά θα πρέπει και να προσπαθούμε βεβαίω να καλύπτονται μια σειρά αποτομή σε αυτέ τι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Αυτό όμως δεν την χάνει της ίδιας υποδοχής από τους εταίρους μας κάθε φορά. Σε κάποιους, ναι, ιδίω ε, από τα μέλη του ΟΣΑ ε, μπορεί να είναι πιο εύκολο να αυξήσει κανείς τον αριθμό των ε, τομέων και των θεμάτων που καλύπτουν αυτέ τι συμφωνίε. Φορολογία, ανταγωνισμό, ακόμη και τέτοια θέματα. Αλλά άμα θέλει κανεί να πάει να μιλήσει με μια λιγότερο ανεπτυγμένη χώρα, και μην πάμε μακριά, ακόμη και με την Ινδία, ένα από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει με την Ινδία και ένα από τα εμπόδια ε, που μας ε, εμποδίζουν στο να συνάψουμε ε, συμφωνία με την Ινδία είναι το ότι η Ινδία θέλει ένα πάρα πολύ χαλαρό κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα. Αδύναμο δηλαδή. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει να μπορεί κανείς και να διαφοροποιεί και να διακρίνει με ποια ε, χώρα κάθε φορά διαπραγματεύεται. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι όλες οι διαδικασίες δεν θα είναι τόσο περίπλοκες, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να καθίστανται εν τέλει ε, ανέφικτες και μη εφαρμόσιμες. Είναι λοιπόν ε, δεδομένο ότι έχουμε πλέον μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες που έχουμε συνάψει τα τελευταία χρόνια και πρέπει καθήκον μας πλέον είναι να αποδείξουμε ότι αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Συμπέρασμά μου λοιπόν είναι ότι αν οι κανόνες είναι υπερβολικά περίπλοκοι, που ούτε καν οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν τις κατανοούν και εδώ πρέπει να αναγνωρίσω ότι η Κομισιόν έχει κάνει αρκετή δουλειά ε, καθήκον μας είναι να τις εξηγήσουμε. Έχουμε πλέον μια στίβα ολόκληρη από σελίδε για το πώς θα εξηγήσουμε τους κανόνες σε μια επιχείρηση. Πώς θα τους εξηγήσουμε ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, να καταγραφούν σε ένα μητρό για να μπορούν να κάνουν εξαγωγές, θα πρέπει να ακολουθούν τον τάδε κανόνα αν θέλουν τα προϊόντα τους να συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο και για τις ίδιες επιχειρήσεις να μπορούν να συμμορφώνονται με αυτές τις συμφωνίες και αυτό είναι εμπόδιο και είναι πρόκληση. Μία λοιπόν από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ότι και εμείς ως επιχειρήσεις θέλουμε οι συμφωνίε αυτές να είναι αποτελεσματικές. Ανησυχούμε. Πράγματι ε, δημιουργούμε ένα σύστημα το οποίο αποφέρει αποτελέσματα πραγματικά ή εν τέλει ε, μιλάμε, μιλάμε, συζητούμε, συζητούμε χωρίς να αποκομίζουμε και τίποτα. Γιατί είναι γεγονό ότι οι δικέ μα διαδικασίε ή οι δικέ μα ε, δομέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ διαφορετικέ από ό,τι στου εταίρου μα. Εμεί έχουμε κοινωνία των πολιτών, κοινωνία των πολιτών. Έχουν όμω όλοι οι εταίροι μα αντίστοιχε δομέ. Πρέπει να κανονίσουμε ότι υπάρχουν διαφορέ λοιπόν. Και δεν μπορούμε απλά να λέμε εντάξει, συνάψαμε τη συμφωνία, σε ένα-δύο μήνε τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται. Όχι. Πρόκειται για μια διαδικασία εν εξελίξη. Ένα, μια δουλειά που θα συνεχίζεται επιμακρών, αν θέλετε. Στόχο μα σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι να συνάψουμε όσο το δυνατόν περισσότερε συμφωνίε οι οποίε θα περιπλέξουν ακόμα περισσότερο του κανόνε. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω το λόγο στου ευρωβουλευτέ ε, όσο το δυνατόν συντομότερα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλύτερη από ποτέ. Συνάπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερε ε, συμφωνίε ε, από το παρελθόν, από ποτεδήποτε, ε, που αποφέρουν και θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση, στην ανάπτυξη. Είναι εμφανή τα απολέγματα. Παλιότερα μιλούσαμε μόνο για ανάπτυξη. Εδώ τώρα πλέον μιλάμε για πολλά θέματα. Εγώ όμω θέλω να φωτίσω μια άλλη διάσταση από αυτή που έχει φωτιστεί από το πάνελ, από του ομιλητέ μα σήμερα. με, δεδομένο, με δεδομένη την στάση των ΗΠΑ, πολλές από τις επιτυχίες μας, όπως με την Ιαπωνία, θα είχαν επιτευχθεί αν δεν είχαν ε, αποσυρθεί οι ΗΠΑ από το TTIP. Θα είχαν επιτευχθεί αν δεν είχαν εξελίξει την ναύτα. Είναι αρκετά καλές οι εμπορικές μας συμφωνίες. Ε, με το Ιαπωνία για παράδειγμα, μετα, μεταφορές δεδομένων, επενδύσεις. Ποιος θα κάνει επενδύσεις. Είμαστε αξιόπιστοι ότι δεν θα επαναληφθούν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με, το, ε, με τον Καναδά. Κάνουμε εν τέλει ό,τι είναι απαραίτητο να κάνουμε για τους ε, κανόνες του εμπορίου. Αξιοποιούμε τον χρόνο και τις συζητήσεις μας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, οι επιτυχίε μα είναι, είναι. Οι επιτυχίε μα μήπω τελικά οφείλονται στι αποτυχίε των άλλων. Κάνουμε πράγματι ό,τι περνά από το χέρι μα για να συνάψουμε εξαιρετικά καλέ εμπορικέ συμφωνίε. Θέλετε να απαντήσετε, κυρία Μάλστρομ. Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς αυτό το ερώτημα βεβαίως. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι είχε ε, κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα το να, το να πει ο, το ότι είπε ο Τραμπ ότι το εμπόριο είναι κακό ή μάλλον είναι καλό όταν με ωφελεί, κακό όταν ωφελεί άλλους. Θετικό ήταν αυτό για να προωθηθούν ε, συμφωνίε οι οποίε είχαν προχωρήσει ήδη αρκετά, όπω με το Μεξικό και την Ιαπωνία. Ήταν σχεδόν έτοιμε να συναυθούν και να, να υπογραφούν, αλλά μπορεί να, να, του έδωσε, έδωσε αυτή η στάση, τον είπα και το, τελικό, την τελική όθηση. Είναι γεγονό ότι ε, το, στο TTP για παράδειγμα ε, είπαν οι χώρες εντάξει είπα εγκαταλείπουν τη διαδικασία ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας υπήρξε λοιπόν μια ωφέλεια ε, για διάφορες πλευρές και κυρίως από την άποψη ότι συνειδητοποιήθηκε και η ανάγκη να, να προστατευτεί και να ε, διαφυλαχθεί το σύστημα του ΠΟΕ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εμείς. Τι να πω, νομίζω ναι. Είναι πάρα πολύ καλές. Μάλλον όχι, γιατί οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες σήμερα πια. Ακόμη και από τότε που δημοσιεύτηκε η αρχική εκδοχή του Trade for All. Ξέρετε, περνάνε πάρα, πολύ, πάρα πολλά στάδια, γιατί δημοσιεύουμε, ανακοινώνουμε, κάνουμε διαβουλεύσεις, μετά περνάμε στη, στη μετάφραση, περνάμε στο κοινοβούλιο, συμβούλιο. Τα πράγματα όμως τρέχουν στο εμπόριο και όταν πλέον ολοκληρώνεται και εγκρίνεται μια στρατηγική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα σε κάποιου τομεί έχουν ήδη αλλάξει. Ελαφρώς μεν, αλλά έχουν αλλάξει. Και ζούμε και σε ένα ψηφιακό κόσμο. Προσπαθούμε συνεχώ. Ναι, όχι λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα οι εμπορικέ συμφωνίε αυτέ δεν είναι αρκετά καλέ. Αλλά άνθρωποι είμαστε. Προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα. Και κυρία Σμικ, ε, συμφωνώ ε, με πολλά από αυτά που είπατε. Αλλά ξέρετε, είναι και ένα θέμα πόρων. Λίγε εκατοντάδε άνθρωποι δουλεύουν στη DG Trade. Είναι ανθρωπίνω ανέφικτο να γίνεται σημαντική πρόοδο σε όλε τι συμφωνίε και σε όλα τα μέτωπα. Σε κάποια σημεία έχουμε ε, προχωρήσει, αλλά ξέρετε, κάποιες, ε, αντιμετωπίζουμε και εμεί κάποιου αντικειμενικούς περιορισμούς ως προς τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας. Um, Θα ακούσουμε μαζί μερικές ερωτήσεις τώρα και μετά την απάντηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να το ε, τοποθετηθώ για κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα που ακούσαμε. Αναφερθήκατε στο Ουσμπεκιστάν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά γιατί καταργήθηκε η παιδική εργασία. Αυτό ισχύει, αλλά υπάρχει καταναγκαστική εργασία πλέον. Αυτό που κάναν παλιά τα παιδιά πλέον το κάνουν ενήλικες μέσω τη καταναγκαστικής εργασία. Όχι ότι κάποιος ε, απειλεί με την απειλή όπλου, με όπλο τους ανθρώπους, αλλά ε, τους αρνούνται τη μισθοδοσία τους αν δεν εργαστούν. Και θέλω να αναφερθώ και σε άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυτική Σαχάρα. Εδώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ε, συγκεκριμένοποιήσει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψη στην προτινόμενη συμφωνία. Αναφέρεται, για παράδειγμα, εκεί ότι οι Ζαράβοι θα πρέπει να ωφεληθούν από την εμπορική συμφωνία. Οι εταιρείε όμως που δραστηριοποιούνται εκεί ε, ανήκουν αποκλειστικά σε Μαροκινούς, επίκους και όχι από Ζαράβη. Άρα η, ο πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας δεν έχει ωφεληθεί καθόλου. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους. Δεν, δεν τους διαβουλεύτηκε κανείς, ούτε καν τους ενημέρωσε. Θιβέτ. ποιο νοιάζεται πια για τέτοιες, ε, τέτοια μικρά και ασήμαντα θέματα όταν έχεις έναν ε, τόσο σημαντικό εταίρο όπως είναι η Κίνα. Αφρική. Τα γεωργικά μας προϊόντα επιδοτούνται σε πολύ σημαντικό βαθμό. Είναι το, τα, μεγαλ, τα περισσότερα κονδύλια της, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατευθύνονται στη γεωργία. Μα καταστρέφουμε όμως την αφρικανική γεωργία με αυτόν τον τρόπο δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε κτηνοτροφία για παράδειγμα έχουν καταστραφεί, έχουν ε, καταργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω ε, των εξαγωγών ε, κρέατος της Ευρώπης στην Αφρική. Αντίστοιχες εξελίξεις είχαμε και στον τομέα του γάλακτος. Η μη επιβολή δασμών εμποδίζει τη δημιουργία εγχώριων βιομηχανιών αυτό σημαίνει ότι είμαστε κι εμεί συνυπεύθυνοι εξαιτία τη εμπορική μα πολιτική για τη συνεχιζόμενη φτώχεια πολλών Αφρικανικών χωρών. Σα ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you very much. Και εμεί ευχαριστούμε. Άντρο και Ευχαριστώ πολύ. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή αυτή ίντα, συνεχίζουμε να ζητάμε ένα σύστημα ελεύθερου εμπορίου και συνολικές ε, συμφωνίες εμπορικές. Μιλάμε για τις προκλήσεις, τα θετικά, τα αρνητικά. Και εγώ θέλω να φερθώ σε κάτι από όλα αυτά. Πρόκειται για τον ε, μηχανισμό διαιτησίας. Οι τελευταίες πληροφορίες που παίρνουμε είναι ανησυχητικέ. Το screening, έτσι όπως το προτείνεται το 2017, όταν η Γερμανία, η Γαλλία και η Μπενελούξ έστειλαν επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κοινή προσέγγιση απέναντι στις ξένες επενδύσεις. Τώρα η Ιταλία προσπαθεί να παρακάμψει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα κυβέρνηση θέλει επενδύσεις από την Κίνα. Πάρα πολλοί επίσημοι από την Ιταλία πηγαίνουν και επισκέπτονται την Κίνα περισσότερες από τις μισές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 13 από τις 28 έχουν ε, μηχανισμούς screening και χώρες όπως η Ιταλία προσπαθούν να παρακάμψουν τους μηχανισμούς αυτούς. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, στην ενιαία αγορά δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά επενδύσεις που έρχονται από τρίτες ε, χώρες, κυρίως από κρατικές επιχειρήσεις και προγράμματα, σε στρατηγικές επενδύσεις και τεχνολογία, δεν είναι φυσιολογικό. Όταν λοιπόν μια κρατική επιχείρηση αποκτά πλήρη έλεγχο της Power Grid στην Πορτογαλία ή 10% των ευρωπαϊκών λιμανιών ε, ελέγχονται από την Κίνα, ή επίση το Ρότερνταμ και την Ανδέρσα έχουν μεγάλα ποσοστά. Τι θα γίνει. Πειραιά, για παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τα πράγματα έτσι. Συνεπώς, κύριε Επίτροπε, ρωτάω. Ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων και ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο όσον αφορά τον μηχανισμό screening για τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Θα υπάρξει συμφωνία μέχρι τα τέλη αυτής της θητείας. Ευχαριστώ. Η κυρία Μινέρ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συντονιστά. Ναι, βάλτε τα ακουστικά σας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθώ τη συζήτηση και τους ομιλητές και τους ευχαριστώ. Ακούω τη Λίνα Κάρκια παράδειγμα, αρκετά ισχυρή κριτική για το πώς προχωράμε και για τις διάφορες ευκαιρίες που έχουμε χάσει, κάτι το οποίο μάλιστα επιβεβαιώνονται και από, από κάποιους από τους άλλους ε, ομιλητές. Η κυρία Μάστρομ λέει ότι αν δεν μπορείτε να τηρήσετε τους κανόνες δεν έχουν νόημα. Ωραία. Το λέει αυτό για τη διαιτησία κυρία Μάλστρομ, αλλά θα έπρεπε να ισχύει και όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις προδιαγραφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες κλπ. που πρέπει να εφαρμόζονται σε τέτοιες συμφωνίες, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Και όμως έτσι επιδεινώνεται το κλίμα με το να μην τηρούνται διάφορες συμφωνίες ή να γίνονται μέσα σε κλειστούς κύκλους, δεν βοηθάμε. Καταστρέφεται ακόμα περισσότερο το περιβάλλον από τις συμφωνίες που γίνονται για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κλπ. Τέτοια πράγματα θα έπρεπε να γίνονται γνωστά. Μιλάμε για το πρόγραμμα Trade for All, εμπόριο για όλους. Δεν ισχύει όμως, γιατί τελικά βοηθούνται περισσότερο μια χούφτα πολυεθνικές. Μα δεν είναι αυτές που χρειάζονται την βοήθεια. Αυτές έχουν μηχανισμό για να διέπουν την οικονομία. Αντίθετα, τη βοήθειά μας πρέπει να τη δίνουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα είπε η κυρία Σάντος. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη στρατηγική ώστε να υποφεληθούν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ε, οι άνθρωποι, τα ζώα, το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν και ρωτάω πότε η εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι πραγματικά για ένα εμπόριο για όλους. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Να υπάρξει επίσης, να προχωρήσει και η υπόθεση της διαιτησίας όσον αφορά την προστασία των διεθνών επενδυτών. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να ενημερώνεται και να έχει λόγο γι' αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και η κυρία Αρενά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Στην ε, σημερινή συζήτηση εκπλήσωμε για την πολιτική μας ανικανότητα να συνειδητοποιήσουμε πόσο πολύ επήγει το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Σίγουρα εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να λύσουν τα πάντα, αλλά ας δίναμε περισσότερη ε, σημασία γιατί το εμπόριο επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή. Η επιτάχυνση του εμπορίου δηλαδή που δεν είναι καλά ρυθμισμένο επιταχύνει τις αρνητικές ε, συνέπειες στο κλίμα. Την κλιματική αλλαγή δηλαδή. Αναρωτιόμαστε συχνά για τις agri-business και πώς η εντατική γεωργία επηρεάζει το κλίμα αρνητικά. Μα φτωχαίνει αποθρεπτικά συστατικά το χώμα. Παρόλα αυτά κάνουμε εμπορικές συμφωνίες εντατικής γεωργίας. Το ίδιο και για την ε, βιοπικιλότητα στη θάλασσα και στη γη. Υπάρχουν ε, Τραγικέ συνέπειε στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, επιταχύνουμε τις εμπορικές μας συναλλαγές με εντατική αλεία. Το ίδιο και για την ε, αποψήλωση. Η Ιαπωνία, η συμφωνία με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφέ προστασίες για τα δάση όπως έχει η Ευρώπη και αυτό που γίνεται στην Ιαπωνία είναι ότι εκεί νομιμοποιείται η συναλλαγή για παράνομη ξυλία. Έπειτα κοινωνικές προδιαγραφές για τους εργαζόμενους. Παράγουμε εκεί που τελικά προστατεύονται λιγότερο οι εργαζόμενοι. Συνεπώς δημιουργούμε έναν αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων. Αυτή είναι η λογική που ακολουθούμε. Οπότε το θέμα δεν είναι να πούμε αν είμαστε για τις ελεύθερες συναλλαγές ή τον προστατευτισμό. Όχι. Αλλά τα εργαλεία ε, οι συμφωνίες αυτές ελεύθερων συναλλαγών μας βοηθούν να αναθεωρήσουμε κάποια λανθασμένα πρότυπα ή αντίθετα πρόκειται για πρότυπα που μας οδηγούν κατευθείαν με το κεφάλι στον τοίχο. Ο συντονιστής, πολλές ήταν οι ερωτήσεις. Θα δώσω στην Επίτροπο βέβαια το λόγο μετά. Ε, αναφερθήκατε στην εφαρμογή στην πράξη και ότι πολύ περισσότερο σήμερα έχουμε να κάνουμε το θέμα της εφαρμογής στην πράξη των συμφωνιών και όχι τόσο με τις διαπραγματεύσεις τους. Η άποψή σας ποια είναι για την ικανότητά μας να εφαρμόσουμε στην πράξη αυτές τις συμφωνίες έτσι όπως τις έχουμε διαπραγματευτεί. Τι λέτε, ο κύριος Μπαρτέλ. Όσον αφορά τη στρατηγική για την εφαρμογή των εμπορικών μας συμφωνιών, ναι, το εμπορικό σκέλος εφαρμόζεται πάρα πολύ καλά, λιγότερο τα εργασιακά και τα περιβαλλοντικά όμως. Μονομερός θα πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εκεί μπαίνουν και τα εργασιακά βέβαια. Υπάρχουν ρήτρε και πολιτικές ε, ρήτρε ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που όμως δεν προχωράνε πάντα εξίσου. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει συγκεκριμένες διατάξεις για να λειτουργήσει κάτι. Από τις εκατοντάδες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που έχουμε, οι περιπτώσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια είναι κάποιες περιπτώσεις ναύτα, ελάχιστες. Δεν σημαίνει ότι δεν παίζει ρόλο το σκέλος της εφαρμογής καθόλου. Αν πάντως η εφαρμογή στον ΠΟΕ αποδυναμωθεί, που είναι μια δυνατότητα, ε, τότε η εφαρμογή των συμφωνιών αυτών θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο βάρος. Πάντως, γενικά μιλώντας, να πω κάτι πολύ σύντομα στο τελευταίο που πήρε το λόγο, αλλά και στους προηγούμενους. Πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στην χρήση μιας εμπορικής συμφωνίας σαν μια μεζούρα που θα κάνει άλλες χώρες να καταλάβουν ότι αν δεν ιτερούν τις υποχρεώσεις τους θα υπάρχουν κυρώσεις ή ε, εξάντερεσιμότητα. Όμως δεν υπάρχει, γιατί η μεζούρα αυτή χρησιμοποιείται για προϊόντα τα οποία δεν είναι απαραίτητα εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται με τον τρόπο ο οποίος δεν μας ικανοποιεί. Από την άλλη, αν συγκρίνουμε αυτό το εργαλείο με ένα εργαλείο περιορισμού της αγοράς σας για τα προϊόντα τα οποία ε, παράγονται με τρόπο που δεν σας ικανοποιεί, αυτό μπορεί να αλλάξει περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή, πρέπει να συνδέονται τα οικονομικά ωφέλη με την παραβίαση τέτοιων προδιαγραφών. Έτσι οι άλλες χώρες θα πιστούν να τηρήσουν τις προδιαγραφές που προσπαθούν να τις κρατήσουν χωριστά από τις συμφωνίες. Η Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχουμε χρόνο να ακούσουμε ερωτήσεις και από τους ε, φοιτητέ. Θα ήταν καλό να τους ακούσουμε. Λοιπόν, για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, ξέρετε ότι είναι ασύμετρες. Δηλαδή δεν ζητάμε από τις χώρες να ανοίξουν τις αγορές τους όπως ανοίγουμε εμείς τις δικές μας. Και προβλέπεται ένα πολύ μεγάλο μέρος για την ανάπτυξη είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να υποχρεωθούν οι χώρες αυτές να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους, να κάνουν εξαγωγέ προ εμά, να δημιουργήσουν υπηρεσίες ασφάλεια τροφίμων κλπ. Αυτή είναι η διαδικασία που προχωράει. Και βοηθάμε και την περιφερειακή ολοκλήρωση στην Αφρική κυρίως ώστε οι συμφωνίες αυτές εταιρικές σχέσεις να αποτελέσουν την βάση για παρετέρω οργάνωση των αφρικανικών χωρών μεταξύ τους. Τώρα, για τον, ε, το screening. Ξέρουμε ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να έχει κάποια ερωτήματα και αμφιβολίες, αλλά έχουν προχωρήσει πολύ, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Ίσως αύριο να υπάρξει τελευταίος τριμερής διάλογος, αν όχι αύριο πολύ σύντομα και ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συντονισμού και ενημέρωσης. Η τελική απόφαση όμως είναι το χωρών μελών. Η Επιτροπή δεν μπορεί να πει ναι ή όχι σε κάποια επένδυση. Εμείς θέλουμε επενδύσεις, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι διακυδεύεται. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της μιας της άλλης χώρας, οι επενδύσεις μας ενδιαφέρουν. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη. Ναι, κυρώσεις. Αλλά δεν έχουμε κυρώσεις όπως θα ήθελε η κυρία Κάρπου και ξέρει γιατί. γιατί υπάρχουν χώρες μέλη που δεν τις θέλουν τις κυρώσεις αυτές. Και γιατί δεν είμαστε και σίγουροι ότι θα έχουν αποτελέσματα. Κανείς δεν τις έχει χρησιμοποιήσει, οπότε δεν ξέρουμε. Αν υπάρξει κάτι πιο ήπιο, μπορεί να βοηθούσε περισσότερο. Και προσπαθούμε ανάλογα με τις προϋποθέσεις να πιέσουμε τις χώρες να τηρούν τους κανόνες για τα εργασιακά, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ρήτρε στις πολιτικές συμφωνίες με πολλές από αυτές τις χώρες. Και δουλεύει. Μόλις γυρίσαμε από το Περού, κάνουν πράγματα με την κοινωνία των πολιτών που ποτέ νωρίτερα δεν είχα φανταστεί ότι θα κάνανε. Χρειάζεται χρόνος με την Κολοβία, τη Γεωργία, οι γυναίκες στην κοινωνία των πολιτών συμμετέχουν, κάτι που δεν γινόταν παλιά. Οπότε δημιουργούν οι συμφωνίες αυτές οι εμπορικές και επενδύσεις και θέσεις ε, εργασίας και η Πορτογαλία για παράδειγμα βοηθήθηκε πάρα πολύ να βγει από την οικονομική κρίση. Δεν είναι το μόνο εργαλείο, συνεισφέρει όμως και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που υπόθηκε πριν ότι πρέπει να επικεντρώμαστε περισσότερο σε αυτούς που χάνουν το δρόμο. Τους πάντα μου αρέσει πολύ αυτή η έκφραση, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το συζητάμε και εδώ το έχουμε συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τις χώρες μέλη. Πριν βρεθούμε σε νέα κρίση, πώς θα επικεντρωθούμε στην ε, συμμετοχή όλων, στην εκπαίδευση, γιατί πολλοί άνθρωποι βρεθήκαν να παίξουν αλήθεια πριν η πραγματικότητα μας ξαναχτυπήσει. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ναι. Οι φοιτητές έχουν ετοιμάσει ερωτήσεις, είναι αλήθεια. Οπότε, σύντομα παρακαλώ με τις ερωτήσεις σας. Σάρλι Κάβεν. Είμαι στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν. Μα είπατε για το σύστημα πολυμερών διαπραγματεύσεων, των ΠΟΕ και τη δράση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά της Κίνας ε, για τι παραβιάσει IP. Ε, η πολιτική Trade for All ε, συζητά τι υπεύθυνε εμπορικέ δράσει και οι αξίε εδώ είναι κεντρική σημασία, όπω η μόρφωση με το σύστημα κανόνων που ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηρίξει το σύστημα αυτό και να εξυπηρετήσει την επίλυση διαφορών και το σχετικό σώμα του ΠΟΕ, εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση. Πόσο είναι σε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως ο ΠΟΕ, για να αντιμετωπίσει την έλλειψη συμμόρφωση τη Κίνας, ε, προκειμένου. Γεια σας. Λέγομαι Στεφάνο και με την κυρία Στατίνη εκπροσωπούμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών. Η ερώτησή μου είναι εξή. Ξέρουμε ότι η κυρία Μάνστρομ ζητά περισσότερη υπευθυνότητα για την διεξαγωγή εμπορικών συμφωνιών και τη σύναψή τους και ξέρουμε τι υπόθηκε στις συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο Γιούνκερ. σε αυτό το στάδιο του εμπορικού πολέμου Ευρωπαϊκή Ένωση είπα. Τι έχετε σκοπό να κάνετε, θα υπάρξουν αντίπεινα ε, επειδή μπορεί να επιβληθούν δασμοί στα εμπορικά αγαθά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε σκοπό να αναλάβετε δράση για να ε, αποκαταστήσετε τις σχέσεις των δύο μερών. Ε, προστατευτισμός μας απειλεί ή λαϊκισμός και είναι τελικά οι δασμοί ένα μέσο για να ασκηθεί πίεση. Ευχαριστούμε. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα τα συνδυαζούμε. Θα συνδυάσουμε με τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Ο κύριος... Επειδή είπατε ότι έχετε βάλει το χρονόμετρο για να δούμε μέχρι πότε θα αναφερθεί το Brexit, εγώ ε, βάζω το χρονόμετρο για να δω πότε θα πρωταναφερθούν οι, μικρο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 50 λεπτά πέρασαν και το είπε η κυρία Σάντος και στο 47 επίσης στο 74 μάλλον, το ανέφερε η κυρία Σάντος. ήταν ε, ένα σοβαρό ερώτημα το κατά πόσο μπορούν οι μικρομεσαίες να αξιοποιήσουν τις εμπορικές μας συμφωνίες. Εάν έχουν πρόσβαση, αν έχουν αρκετές πληροφορίες, αν υπάρχουν ε, γλωσσικοί φραγμοί ε, μπορεί να εμποδίζουν τις μικρομεσαίες οι γλωσσικοί περιορισμοί. Δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα. Πού υπάρχει λοιπόν δυνατότητα να γίνουν πιο αποτελεσματικέ εμπορικέ μα συμφωνίε. Ναι, πιστεύω, αν και μπορεί να κάνω λάθο, ότι 90% του χρόνου συζητάμε για τη δυνατότητά μα να εξάγουμε πρότυπα και αξίε μέσω των συμφωνίων ελεύθερου εμπορίου. Μήπω συζητάμε και λίγο για τη δυνατότητά μα να εξάγουμε αγαθάκια υπηρεσίε, διότι τελικά οι εμπορικέ συμφωνίε αυτό θα έπρεπε να αφορούν. Την εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Άμα δεν τα πάνε καλά οι εταιρείε και επιχειρήσει, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει μα, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα υπόλοιπα, τίποτα. Δεν λέω ότι τα άλλα ζητήματα που περιμένουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ε, δεν είναι ε, καλά. Αλλά εμπορικέ συμφωνίε άλλο ε, στόχο έχουν ποτίστω. Και νομίζω και εσεί, Επίτροπε, πολύ σωστά τα αναφέρατε στην αρχή αυτά που είναι ζωτική σημασία και το κατά πόσο πρέπει να υπάρξει σωστή κατανομή των ωφελών τη παγκοσμιοποίηση. Αλλά πρώτα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οι μικρομεσαίες της Ανατολής και της Δύσης να εφηληθούν εξίσου. Εάν συγκρίνετε την Πορτογαλία με τη Ρουμανία στις μικρομεσαίες τους ή τη Φιλανδία και τη Σουηδία ας πούμε, ε, το χάσμα είναι τεράστιο. Δεν έχω λοιπόν ερώτηση, αλλά μια παρατήρηση. Σήμερα αυτή η εμπορική πολιτική μου φαίνεται ότι έχει γίνει ένα χρησιμότατο εργαλείο για να έχουμε και μια εμπορική πολιτική και μια πολιτική εργασία και ημέρα συζήτηση τη πολιτική εργασία στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Αφού συζητούμε το τι υπόθηκε προηγουμένω, να συζητήσω κι εγώ κάποια από αυτά που υπόθηκαν πριν, από τα σχόλια της κυρίας Σάντο. Βεβαίω πρέπει να προωθήσουμε το εμπόριο, αλλά δεν μπορεί και η εμπορική πολιτική μόνη τη να λύσει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του κόσμου. Πολύ σημαντική παρατήρηση αυτή που κάνατε. Όμω είναι και δική μα υποχρέωση να προωθήσουμε τι αξίε μα εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνία, Συμφωνία Εταιρική Οικονομική Σχέση. Η Ιαπωνία πρωτού γκρίνει την ε, συμφωνία έλαβε μέτρα για την αποκομιδή των ε, αποβλήτων στη θάλασσα. Ήδη από το G7 το είχε υποσχεθεί στην Οζάκα για το G20 του χρόνου. Είναι ήδη κάτι αυτό. Βλέπουμε ότι έχουν κάποιο αντίκτυπο εμπορικέ συμφωνίε και είναι σημαντικό να το λέμε. Επ' αυτού είμαι σκιώδης εισηγητή του ΕΛΚ συγκεκριμένα. Γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Και το έβαλε στο Twitter και έλαβα πάρα πολλά σχόλια χιονοστιβάδα, αλλά μου πάνε μεγάλε εταιρείε μόνο ωφελούνται. Και είπα, ναι, ε, λογικό είναι μεγάλοι να ωφεληθούν πρώτοι. Αλλά έχουμε ειδικό κεφάλαιο για του μικρομεσαίε και είναι και αυτό σημαντικό. Και με ξαναρώτησαν τι οικονομικό κέρδο θα έχουμε. Τι είναι 0,0 κάτι του ΑΕΠ. Και εγώ είπα ότι ναι, μπορεί να φαίνεται πολύ μικρό το ποσό, Όμω, με την καλλιέργεια και τη δημιουργία οικονομικού κέρδους δημιουργούμε και θέσεις εργασία και αυτό μας μοιάζει. Εκεί είναι η κοινωνική πρόοδο. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά. Τι εμπορικού εταίρους ψάχνουμε. Διότι ο ιδανικός εμπορικός εταίρος δεν υπάρχει. Κανείς δεν είναι τέλειο. Ακόμη και αν πάτε σε γειτονικέ ευρωπαϊκέ χώρε, θα δείτε ότι κάποιοι δεν σέβονται πλήρω το κάτω δικαίου. Άλλοι δεν σέβονται πλήρω κάτι άλλο. Οπότε δεν μπορούμε να βρούμε κανένα που να είναι ο τέλειο μαθητή. Και τελευταία παρατήρηση για τη διαφάνεια. Και εδώ το θέτω προ του φοιτητέ μα. Διότι η διαφάνεια έχει βελτιωθεί, έχει αυξηθεί. Τώρα μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίε για τι διεξαγωγή διαπραγματεύσει εγκαίρω. Την περασμένη εβδομάδα όμω είχαμε μια συνάντηση ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο και ένα από αυτού ρωτούσε το εξή. Άλλα έγγραφα δεν υπάρχουν διαθέσιμα για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνία. Ναι, από πέρσι το Δεκέμβριο. Αλλά ο κύριο Ευρωβουλευτή δεν ήξερε πού να πάει να τα βρει. Δεν είχε ενημερωθεί αναλόγω. Να ένα πρόβλημα λοιπόν. Πρέπει να σκεφτούμε πώς εσείς, εσείς πρέπει να προωθήσετε τα ωφέλη αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Εσείς τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να τα γνωρίζετε καλύτερα την ερώτηση προς σας. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Πινιέρο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους όσοι πήρατε το λόγο. Είναι μια συζήτηση με πολύ περιεχόμενο. Πραγματικά άξιζε τον κόπο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι μισογεμάτο το ποτήρι. Όντως προχωρήσαμε πολύ σε θέματα κοινωνικά, σε θέματα εμπορικών κύκλων. Οι προοπτικές έχουν βελτιωθεί. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα νομίζω ότι υπάρχουν δύο πολύ καλές ρυθμίσεις που ξεχνάμε συχνά. Είναι εκείνες που έχουν να κάνουν με την εξοριστική βιομηχανία εκεί όπου υπάρχουν συγκρούσεις και το θέμα της θανατικής ποινής. Αυτά τα δύο πρέπει να τα προβάλλουμε. Φυσικά παραμένουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα, να βελτιωθούν τόσο όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά όσον αφορά και την εφαρμογή στην πράξη των συμφωνιών. Τώρα, σε σχέση με το όσα άκουσα εδώ, η εμπορική πολιτική αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο από πλευρά γεωστρατηγικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δύσκολα μπορεί να βαρύνει στη διεθνή σκηνή αν δεν έχει οικονομικό βάρος. Πρέπει να το έχουμε. Συνεπώς πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι η Κίνα τα τελευταία 15 χρόνια έχει γίνει η δεύτερη παγκόσμια δύναμη και έχει προσπεράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτού. Οι Ηνωμένε Πολιτείε εξακολουθούν να είναι η πρώτη παγκόσμια δύναμη, όμως η απόσταση όσον αφορά το βάρος ε, της ε, κάθε οικονομίας σε σχέση με το ΕΠ έχει μειωθεί μόνο κατά 9 μονάδες. Απ' την άλλη υπάρχει η στρατηγική οικονομική του Τραμπ που θέλει να επαναφέρει τη χώρα με το America First που στην πραγματικότητα δεν θέλει να είναι America First, θέλει να είναι America Only. Οπότε η στρατηγική του είναι πολύ συγκεκριμένη. Μια προστατευτική εμπορική πολιτική υπέρ των συμφερόντων των ΗΠΑ με μια ε, χρηματοπιστωτική και φορολογική πολιτική τέτοια ώστε να επιστρέψουν οι επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήθελα να έχουμε μια συνολική στρατηγική για τα γεωπολιτικά μας. Ας πούμε να είχαμε περισσότερα μέσα και πόρους στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Εδώ η δικιά μας Επιτροπή πάντα ζητάει με τροπολογία αύξηση των πόρων. Γιατί δεν θέλουμε να παραμένουμε με συμφωνίες που έχουν ξεπεραστεί από το χρόνο. Χρειαζόμαστε καλύτερη στρατηγική λοιπόν σε σχέση με τη βιομηχανική πολιτική, την ενεργειακή, υποδομών, μεταφορών, γιατί μόνο τότε μπορείς να είσαι πραγματικά ανταγωνιστικός και έτσι να βαραίνει περισσότερο η θέση σου στη στρατηγική που θα προτείνεις. και αυτοί που έχουν να κερδίσουν είναι ακριβώς αυτοί των οποίων το βάρος είναι πιο μεγάλο. Αυτοί γίνονται σεβαστοί από την παγκόσμια σκηνή. Τίποτα άλλο. Η Επίτροπος. Οι περισσότερες ερωτήσεις απευθύνθηκαν σε μένα. Ο κύριος πρώτα ή όχι. Όχι, εσείς κάνατε την πρώτη ερώτηση. Δεν μπορεί ποτέ ε, να είναι βέβαιο για το τι θα αποφασίσει ο ΠΟΕ, αλλά πριν προσφύγουμε κατά οποιασδήποτε χώρα στον ΠΟΕ, έχουμε πολύ διεξοδική νομική εξέταση του θέματος για να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε κάνει ήδη το σωστό. Το πρόβλημα με τον ΠΟΕ αυτή τη στιγμή είναι ότι το αρμόδιο σώμα θα ε, πεθάνει Εάν δεν γίνει τίποτα του χρόνου, θα πάψει να λειτουργεί. Εάν λοιπόν πάμε πρωτοβαθμίω, οπότε αν εδώ ρωτάτε για την Κίνα ή για οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση, αν δεν υπάρχει σχετικό σώμα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Κοιτάζουμε λοιπόν τώρα να συγκεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα για να δούμε πώ μπορούμε να σώσουμε το αρμόδιο σώμα του ΠΟΕ, αλλά δεν έχουμε και επίκαιρου κανόνε, επικαιροποιημένου κανόνε των ΠΟΕ. Κατηγορούμε την Κίνα για πολλά πράγματα, αλλά δεν αναφέρονται πουθενά στου κανόνε, στην ε, μεταβολή τη τεχνολογία, και το κ.ο.κ. Αυτά έχουμε αρχίσει με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία να τα να βάλουμε σε ένα κείμενο, να υποβάλουμε κάποια πρόταση για να αναλάβει ο καθένα και τι ευθύνε του, συγκεκριμένα η Κίνα. Ιδάλω, ε, ο ΠΟΕ γίνεται λιγάκι απαρχιωμένο, πράγμα που ήδη συμβαίνει σήμερα σε έναν βαθμό. Για την άλλη σα ερώτηση, ένα, εάν οι υπάρχει να επιβάλλουν δασμού για τα ανταλλακτικά αυτοκίνητα κάτι που δεν νομίζουμε θα κάνουμε, διότι θα ήταν αδικαιολόγητο. Ναι, θα λαμβάναμε αντίμετρα. Δεν θέλουμε, διότι τότε υπάρχει κλιμάκωση. Όμω, είναι τελείω παράνομο να αναλάβει κανεί τέτοια δράση. Δεν μπορεί να λέει κανεί ότι οι εξαγωγέ αυτοκινήτων ε, προ τι τι ΗΠΑ δημιουργούν ε, κίνδυνο δημόσια ασφάλεια. και είμαστε και σε πλήρη συμμόρφωση με του κανόνε του ΠΟΕ. Ε, μπορούμε να υπολογίσουμε κατά λεπτό στο τι έχει συμβεί. Και βεβαίω θα το κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω θα προχωρήσει με την πλήρη συμφωνία των 100 μελών και θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Για τι μικρομεσαίε, κύριε Βίνκλε, συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Το ανέφερα στην ομιλία μου, αλλά δεν έχουμε δώσει τι προσοχή Πολύ περισσότερα μπορούν να γίνουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα κεφάλαια για αυτό. Ε, με σημεία επαφή σε κάθε χώρα προσπαθούμε να τα δημιουργήσουμε. Προσπαθούμε να έχουμε επαφή με τα επιμελητήρια των μικρομεσαίων στι διάφορε χώρε. Συνεργαζόμαστε με την Business Europe, ε, με την Ένωση των Μικρομεσαίων δηλαδή. Αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, διευκόλυνση με φιλικότερα προς το χρήστη site. Ναι, Σίγουρα πολλά μπορούν να γίνουν τι μικρομεσαίε. Σε συνεργασία με τι επιχειρήσει στα για να διαδοθεί η γνώση που διαθέτουμε, να ενθαρρύνουμε αυτού που θέλουν να ε, πάνε για εμπόριο στο εξωτερικό να το κάνουν. Βεβαίω χρειάζονται στήριξη και μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και για την ερώτηση τη ΣΥΜΑ. Προσπαθούμε να έχουμε μια ε, συνεκτική στρατηγική ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το εμπόριο, την περιβάλλον, την εργασία, ό,τι μπορούμε με τις χώρες μέλη μας. Κάποιες είναι στρατηγικοί εταίροι. Κάποιες χρειάζονται μια συνολικότερη στρατηγική, γιατί έχουμε πιο μακροπρόθεσμους στόχους είναι εταίρος και σε άλλους τομείς. Άλλοι πρέπει να προχωρήσουν στην ανάπτυξή τους, όμως ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους συναδέλφους μου. Και σίγουρα και πάλι υπάρχει περιθώριο να τα πάμε και καλύτερα. In addition, yes, we support. Να προσθέσω κι εγώ ότι εμείς ε, υποστηρίζουμε βεβαίως τις ε, κινήσεις σας, τους τρεις πυλώνες, τα αντίμετρα που στόχο έχουν να προφυλάξουν και να διαφυλάξουν τον ε, ΠΟΕ και, την, ε, και τις αγορές. Είναι σαφές ότι εμείς ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και είμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν ο Καναδάς και το Μεξικό. Για μας είναι ξεκάθαρο. Η απάντηση στο πρώτα η Αμερική είναι ενωμένη η Ευρώπη. Ναι. Θέλω να πω και εγώ κάποια πράγματα, απαντώντας στα όσα είπε η κυρία Μάλστρομ όσον αφορά τους περιορισμένους πόρους για την παρακολούθηση. Όλοι το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Αλλά ένας σχετικά απλό τρόπος για να ε, βελτιώσει κανείς την παρακολούθηση και την επιβολή των συμφωνιών είναι να δοθεί ένας μηχανισμός στους εμπλεκόμενους, στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να μπορούν να κοινοποιούν πληροφορίες ή να υποβάλουν αιτήματα ώστε να μην χρειάζεται να πας εσύ να τους βρεις, αλλά τα ίδια τα ζητήματα να έρχονται να βρίσκουν εσένα από τους εμπλεκόμενους για τις κυρώσεις. Το συζητάμε εδώ και τρία χρόνια. Κανείς δεν, έχει, επιβάλει ποτέ, δεν ξέρουμε αν είναι αποτελεσματική. Αλλά όσο ακόμα συζητούνταν το TTIP, υπήρξε μια συζήτηση με τους ε, για τα εργασιακά διαπραγματευτές και εκείνος μας είπε ότι το σύστημα των ΙΠΑ και το σύστημα κυρώσεων που έχουν για τα εργασιακά ε, μας είπε λοιπόν ότι αν δεν υπάρχουν κυρώσεις, ποιος θα μας πάρει στα σοβαρά δεν είναι απαραίτητο να τις επιβάλλεις με, με την πρώτη ευκαιρία. Αλλά σε τελική ανάλυση πρόκειται για ένα μηχανισμό που σε κάνει πιο αξιόπιστο στα μάτια του εταίρου σου. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός επιβολής κυρώσεων. Όταν μιλάμε για τα ποτήρια που είναι μισοάδια ή μισογεμάτα, μπορεί ε, τα, οι δικέ μου παρατηρήσει να ακούστηκαν αρνητικέ. Αλλά πρέπει να σα πω ότι και εγώ αισιόδοξη είμαι. Φυσικά και το εμπόριο δεν μπορεί να λύσει τα πάντα, όλα τα προβλήματα. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι πλέον υπάρχει και το θεματολόγιο του, του ΟΗΕ για το 2030 και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εκεί περιλαμβάνονται μια σειρά από ζητήματα που αφορούν και εμά, αφορούν και του εταίρου μα, είτε είναι ανεπτυγμένοι είτε λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε. Και όταν κάνουμε διαπραγματεύσει για τέτοιε συμφωνίε ελευθερών συναλλαγών θα πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι το εμπόριο το οποίο επιδιώκουμε θα πρέπει να είναι ένα εμπόριο δίκαιο που θα βασίζεται σε κανόνες, που θα σέβεται τα εργατικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα το περιβάλλον και που θα προάγει τα δικαιώματα αυτά και δεν θα τα καταπατά. Να κάνω μια ερώτηση για αυτά που είπατε για τα εργασιακά Είπα πρόσφατα ε, υπερέβησαν στην αυτά το ζήτημα της εξάντε αιρεσιμότητας και μάλιστα ε, συμπεριέλαβαν πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Μέχρι και 16 δολάρια την ώρα είπαν. Ε, είναι και αυτό ένα μέσο. Εσείς θα συμφανούσατε ή όχι. Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου αυτή που μου θέτεται αν γραμματικά κάποιος μπορεί να καταλάβει τι προτείνουν οι ΙΠΑ. Διότι εμείς μιλάμε με τους συναδέλφους μας από τις ΙΠΑ, με τα συνδικάτα και του ρωτάμε τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα, μπορείτε να μας εξηγήσετε, τι, τι εννοούν, τι επιδιώκουν με αυτή την απέτηση. Ένα συγκεκριμένο ποσοστό δηλαδή του παραγόμενου πλούτου θα να πρέπει να παράγεται από εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με συγκεκριμένο ορομίστιο. Κανείς δεν είναι σε θέση να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Και είναι σαφές ότι στο σύγχρονο κόσμο τα αγαθά δεν παράγονται πλέον σε ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο. Υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα και τμήματα ενός προϊόντος το οποίο μπορεί να έχουν παραχθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου. Άρα μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει συμμόρφωση με αυτή την απέτηση αν κατά την παραγωγή των εξαρτημάτων υπήρξε, ε, ε, τηρούνταν αυτό ο κανόνα, αλλά μπορεί να μην υπάρχει συμμόρφωση αν τα εξαρτήματα αυτά έχουν συναρμολογηθεί στο Μεξικό. Δεν ξέρει κανεί τι συμβαίνει. Όχι για αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά αυτό που βλέπουμε με τον ILO είναι ότι ε, ε, συνεργαζόμαστε στην περίπτωση της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα υπήρχαν κυρώσεις στο Μεξικό και στον Καναδά θα υπήρχαν όσον αφορά τις εργασιακές διατάξεις δικός μας στόχος και καθήκον είναι να συνδράμουμε τεχνικά να μακροπρόθεσμα γιατί όλα αυτά αφορούν και την τροποποίηση νομοθεσίας που ισχύει σε μια χώρα ε, μιλάμε για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον, μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, ε, προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, παροχή της δυνατότητας σε αυτές να μπορούν να επιτύχουν τους στόχους. Δεν έχουμε εμείς συγκεκριμένη θέση για το αν οι είναι καλό πράγμα ή κακό. Εμείς καλούμαστε και ανταποκρινόμαστε σε κάθε περίπτωση είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν. Στόχος μας είναι αυτή η μακροπρόθεσμη οι μακροπρόθεσμες στοχεύσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση εμπιστοσύνη και για την επίτευξη του στόχου αξιοπρεπή εργασία για όλου μακροπρόθεσμα. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον, ε, το εμπόριο, αφορά μια σειρά από τομεί πολιτική, αφορά και την τεχνική συνεργασία και είναι ένα τρόπο για να, να οι ανισότητε, ο κοινωνικό αποκλεισμό κτλ. Συχνά και στους εποπτικούς μας μηχανισμούς πρέπει να σας πω ότι δεν δείχνουμε τα δόντια μας, δεν επιβάλλουμε κυρώσεις. Όταν λαμβάνονται αποφάσεις από τους δικούς μας φορείς, Μπορεί κάποιοι να το εκλαμβάνουν αυτό ω κατηγορητήριο που απευθύνουμε σε συγκεκριμένε χώρε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διακόπτουμε τον διάλογο. Εμεί ω τριμερή οργανισμό. Δεν χάνουμε τον έλεγχο της κατάστασης. Εμένουμε, επιμένουμε στο έργο μας με μακρόπνοη και μακρόχρονη στόχευση. Um, να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Όταν οι δημοκρατικοί κατέκτησαν το, τη γερουσία, άρχισαν να συντάσσουν νομοθεσία, νομοσχέδια δηλαδή, που ε, περιλάμβαναν και πολλά πρότυπα του ε, ILO. Ε, ένα συγκεκριμένα μάλιστα που αφορούσε την εργασία των ε, κρατουμένων. Σε ποιο βαθμό οι συμβάσεις του ILO τελικά αποτελούν όμως εμπόδιο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορείτε να, να, να επαναλάβετε. Στις ΗΠΑ θεωρήθηκε ότι παραβιάζονται τα πρότυπα του ILO μέσω εργασιών του, του, του Κογκρέσου, νομοσχεδίων που κατατέθηκαν εκεί. Όλοι γνωρίζουμε ότι κάποιες από τις πλούσιες χώρες δεν έχουν κυρώσει τις βασικές συμβάσεις και η ΕΠΑ είναι μία από αυτές τις χώρες. Ο Καναδάς επίσης χρειάστηκε πολύ χρόνο μέχρι να κυρώσει όλες τις συμβάσεις του ΑΕΛΟ. Κάποιες φορές είναι κάποια λεπτομέρεια του δικαιικού του συστήματος που τους εμποδίζει να το κάνουν. Ή σε άλλες χώρες υπάρχουν ε, μια σειρά από περιφέρειες που θα πρέπει κάθε μία ξεχωριστά να εγκρίνει του, τις, τις συμβάσεις. Εδώ εμείς παρεμβαίνουμε και συνδράμουμε τις αρχές τεχνικά, αλλά θα πρέπει ως χώρα να είναι κανείς πολύ προσεκτικός ε, όταν θέλει να αναγκάσει μια άλλη χώρα να ακολουθήσει κανόνες στους οποίους η ίδια δεν ακολουθεί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με την οικοδόμηση εμπιστοσύνη ούτε με την έννοια τη αμοιβαιότητα. Αυτό που είδαμε όμω ε, στην έρευνά μα είναι ότι οι συμβάσεις του ILO δεν πλήττουν δυσανάλογα τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Από την έρευνά μας προκύπτει το αντίθετο, και οι φτωχότερες χώρες, αν μου επιτρέπετε να τις πω έτσι, ωφελούνται εν τέλει από το εμπόριο γιατί ενισχύεται η παραγωγικότητα και η συμμετοχή μεγαλύτερου τμήματος του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, αλλά ιδίως γυναικών. Φυσικά, περισσότερα πρέπει να γίνουν να, να διευρυνθεί η έρευνα που έχει γίνει και να στοιχειοθετηθεί και με περισσότερα στοιχεία. Θα έπρεπε να λειτουργεί, να έχει κανείς τα ωφέλη από την νέα ναύτα Οπότε φαίνεται είναι 16 δολάρια την ώρα. Και δεν θέλω να το παρακάνω, αλλά υπάρχει ένα θέμα στρατηγικής. Δηλαδή, πόσο εξάγεις τις δικές σου προδιαγραφές, πώς καταφέρεις άλλες χώρες να, να εφαρμόσουν τις δικές σου προδιαγραφές και μετά πρέπει εσύ να προσαρμόσεις τις δικές σου είναι ένα παλιό πρόβλημα στο εμπορικό δίκαιο. Δηλαδή προωθείς τόσο πολύ τις δικές σου αξίες, το δικό σου σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο ότι θα δυσκολευτούν ένα σωρό επιχειρήσεις να τα βγάλουν πέρα, είναι ότι τελικά βάζεις και έξοδα στους ανταγωνιστές σου. Πώς θα το κάνουνε. Εξού και ο Τραμπ το λέει ότι αν θέλετε να έχετε και πάλι την Αμερική δυνατή, αυτό ακριβώς πρέπει να κάνετε. Ο συντονιστής. Όποτε ταξιδεύω σε αναπτυσσόμενες χώρες και τους ρωτάω για τις εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά ακούω παράπονα για τις προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόσουν οι αγρότες στο Μαλί, για παράδειγμα που μιλάνε, τι μιλάνε, μπαμπάω, έχουν μία λέξη που ήταν τοξίνες που συνέχεια επαναλάμβαναν, γιατί φαίνεται ότι καταστρέφονται οι δικές τους καλλιέργειες εξαιτία των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για τοξίνες στα καρύδια. Και σίγουρα υπάρχει θέμα παζαρέματος του στόχους ασφάλεια, προδιαγραφές, ασφάλεια τροφίμων κλπ. Πρέπει να δούμε πώς θα πετύχουμε την καλύτερη συμφιλίωση. Φαντάζομαι σε αναψώμενες χώρες και εσείς τα ίδια θα έχετε ακούσει που ακούω και εγώ, έτσι δεν είναι. Κατά κάποιο τρόπο ναι, αλλά όχι απαραίτητα. Γιατί θέλω να προσθέσω κι εγώ κάτι που έχει να κάνει με αυτές τις προδιαγραφές. Θέλω να επενθυμίσω για το θέμα της βιωσιμότητας. Έχει τρεις πυλώνες. Και η διεθνής κοινότητα συζήτησε το 2015 τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είπε ότι δεν έχει νόημα να κοιτάμε μόνο έναν πυλώνα. Δεν θα έχουμε ποτέ βιώσιμη ανάπτυξη αν κοιτάμε μόνο την οικονομική πτυχή ή μόνο την κοινωνική ή μόνο το περιβάλλον. Πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη και τα τρία και να έχει πολιτικές συνεπείς και ως προς τους τρεις πυλώνες. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα ότι το σύστημα θα λειτουργήσει μόνο λάβουμε υπόψη μα και τους τρεις πυλώνε, Κάτι το οποίο συχνά ξεχνάμε. Σήμερα δεν μπορεί να πει κάτι όπου υπερφορτώνεις με εμπορικά στοιχεία και όχι με τα κοινωνικά ή το περιβάλλον. Ακριβώς η ιστορία είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάς μόνο έναν από τους τρεις πυλώνες. Πρέπει να τους συνδυάζει και τους τρεις. Και το θέμα των προδιαγραφών φυσικά και είναι δύσκολο. Η συμμόρφωση δηλαδή πολλών αναπτυσσόμενων χωρών. Αλλά αυτό ακριβώς είναι που προσπαθεί να διορθώσει και αναπτυξιακή ε, πολιτική και βοήθεια. Όμως, στις αναπτυσσόμενες χώρες όταν προσπαθούν να βελτιώσουν τις προδιαγραφές, ε, βελτιώνουν την κατάσταση στις χώρες αυτές, γιατί και αυτοί χρειάζονται προστασία των καταναλωτών τους και αυτοί χρειάζονται περιβαλλοντική πολιτική. Οπότε η προσαρμογή τους στις δικές μας ε, τις προδιαγραφές βοηθάει τις δικές τους κοινωνίες. Αλλά είναι το αναπτυξιακό που πρέπει να προσέχουμε. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, μερικές φορές το επιχείρημα που ακούει κανείς είναι ότι οι εκεί πρέπει να συμμαρφώνονται και με δικές μας προδιαγραφές, ας πούμε, των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Όταν πάνε οι προμηθευτές, ε, τους ζητάνε μια ολόκληρη σειρά προδιαγραφών. Θα ήταν πιο εύκολο αν οι χώρες μπορούσαν να δημιουργήσουν τις δικές τους ισχυρές προδιαγραφές. ενώ τώρα επιβάλλουμε. Θα ήταν προς το συμφέρον τους. Οι βιομηχανικές χώρες πρέπει να στηρίξουν τη δημιουργία ε, υποδομών ποιότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ωραία, όταν μιλήσατε για 13 ευρώ την ώρα, έτσι είπατε στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Δεν αναφέρεται ρητά βέβαια. Αλλά τελικά αυτή είναι η τιμή του να κάνει κανείς business με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι είπατε. Ναι, ισχύει αυτό δεν νομίζω ότι θα το συμπεριλάβουμε στις εμπορικές μας συμφωνίες πόσα ευρώ θα πρέπει να πληρώνονται, τουλάχιστον έτσι, τώρα άμεσα. Αλλά επίσης αληθεύει. Δεν έχω πάει στο Μαλί, αλλά και σε άλλες αφρικανικές χώρες έχω ακούσει ανάλογα παραδείγματα και παράπονα. Αυτό έχει να κάνει με τους κανονισμούς των φυτογειονομικών που αφορούν την προστασία των καταναλωτών μας εδώ στην Ευρώπη. Δεν ε, βλέπω γιατί θα έπρεπε να αλλάξουμε κάτι σε αυτό και να υποχωρήσουμε. Πώς θα αποκτούσαμε την εμπιστοσύνη των δικών μας πολιτών. Ε, και οι άλλες χώρες πρέπει να αυξήσουν τη δική τους διατροφική ασφάλεια με τους αρμόδιους φορείς και σώματα εκεί, τους ε, οικίους φορείς και σώματα για δικό τους όφελος Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλο εμπορικό εταίρο. Επιβάλλουμε πολλά πρότυπα, ακόμη και αν τα περισσότερα από αυτά είναι και διεθνή, σε υψηλό βαθμό. Περισσότερο και από, τους, από τη ΣΥΠΑ. Χρησιμοποιούμε περισσότερα διεθνή πρότυπα και εκπονούμε και περισσότερη νομοθεσία. Δεν είναι η πρόθεση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων να γίνει εμπορικό εργαλείο, αλλά είναι μια επίπτωση, συνέπεια που ε, ε, προκύπτει. Ε, έχουν γίνει κάποια παράπονα, αλλά και σε άλλε χώρε προσπαθούν να βρουν το δικό του κανόνα προστασία δεδομένων. Γιατί ναι, πρέπει να βρούμε την προστασία των δεδομένων μεν ω στόχο, αλλά πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με τα προσωπικά δεδομένα. Προσπαθούν να βρουν ένα σημείο ισορροπία. Η Ιαπωνία κάνει τα ανάλογα και άλλε χώρε. Οπότε το εμπόριο προσπαθεί να καλύψει όσα περισσότερα γίνεται, αλλά και να μην τα υπερκαλύπτει. Υπάρχουν ε, πολλοί κανόνες που δεν έχουν σκοπό να καλύψουν εμπορικά ζητήματα πρωταρχικώ. αλλά ίσως να είναι το όριο, όπω είπατε, τα 16 ευρώ. Δεν το βλέπω όμω να γίνεται στο άμεσο μέλλον. Και τα δεδομένα. Τα δεδομένα ήταν ένα ε, ζήτημα αμφιλεγόμενο και εντό Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άκουσα ένα Επιχείρημα που συχνά ακούγεται από τη Γενική Διεύθυνση Trade. Καλύτερα να γράφατε πιο συγκεκριμένου κανόνε στι εμπορικέ συμφωνίε. Ε, είπα το κάνουν. Τουλάχιστον θα κάνουν συνειδητέ επιλογέ μετά οι υπόλοιποι την να εφαρμόσουν. Και θα ξέραμε τι εξάγουμε και τι όχι. Γιατί υπάρχουν ρήτρε για δεδομένα. στις Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που έχουν κάποια ισοδύναμα και αντιστοιχίε που είναι δύσκολο να εξακριβωθούν. Κοιτάξτε, ε, θα συμφωνούσα, αλλά είναι μια, ένα συμβασμό που γίνεται με πολλού εταίρου και έχει, έχει συνέπειες και για το εμπόριο. Σίγουρα είναι κάτι όμω που θα το σκεφτούμε στο μέλλον. Λούση, να σε ρωτήσω για τι επιχειρήσει και την άποψή του γι' αυτό, διότι αυτορμήτω οι επιχειρήσει δεν συμπαθούν τους κανόνες. Όμω άκουσα πολλέ εταιρείε να λένε ότι άμα συμμορφωθεί κανεί με του κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν να έχει τελειώσει με τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτό αν το έχει κανεί στην αγορά του. Άρα είναι μάλλον διευκολυντικό. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να το δει κανείς αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε ατζέντα απορρίθμιση ε, για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Έχουμε ατζέντα καλύτερη νομοθεσία. Και υπάρχει διαφορά. Υπάρχει διαφορά διότι. Να πάω λίγο πίσω σε αυτά που είπα. Δεν είναι το θέμα της ποσότητας κατά της ποιότητας. Αυτό ισχύει και για τις εμπορικές συμφωνίες και για τους κανόνες και τις ρυθμίσεις. Πρέπει να βεβαιωθεί κανεί, ότι είναι αποτελεσματικά είναι σημαντική προκειμένου να πετυχάνουν τους στόχους τους. Συμφωνώ απολύτως ότι ζούμε σε μια κοινωνία όπου έχουμε υψηλά πρότυπα και στα κοινωνικά και στα περιβαλλοντικά και στην προστασία των καταναλωτών και σε όλους αυτούς τους τομείς. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν προσαρμοστεί και θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται και να δημιουργούν την απαραίτητη τεχνολογία και τις τεχνολογικές λύσεις που θα μας επιτρέπουν να εκπληρώνουμε κάποιε από αυτέ τι προποθέσει και αυτού του κανόνε να του τηρούμε. Για τι κλιματικέ αλλαγέ, α πούμε, για την αναχέτηση του αντικτύπου των κλιματικών αλλαγών, πρέπει να γίνει πολλή δουλειά. Πρέπει όμω να γίνει προσπάθεια και από την κοινότητα των επιχειρήσεων και των εταιριών τεχνολογία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Υπάρχουν όμω και κανόνε που δεν επηρεάζουν την κοινότητα. Γιατί Προφανώ το να εκπονούμε κανόνε είναι καλό και για του πολίτε και για την κοινωνία μα, αλλά δεν νομίζουμε ότι αναστέλει τη δυνατότητά μα να ανταγωνιζόμαστε στο εξωτερικό, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε υπέρ με του κανόνε που να το κάνουν αυτό. Δεν είναι υπέρ των καταναλωτών, των, των ε, χρηστών. Ε, δεν υπάρχει λόγο να επιβάλλουμε κανόνε στι εταιρείε και τι επιχειρήσει μα, εάν δεν τι επιτρέπουμε να είναι ανταγωνιστικότεροι και να καινοτομούν. Και στον τομέα των δεδομένων, Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα δεδομένα και τι εμπορικέ συμφωνίε, απέχουμε πολύ από ένα ιδεατό σενάριο και σκηνικό. Είναι ένα τομέα που χρειαζόμαστε περισσότερε προσπάθειες και θα έλεγα ότι το GDPR, αυτό ο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικότατο ο ιδιωτικό βίο, αλλά διαρκώ μα ε, απειλούν επιθέσεις στον χώρο. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα ε, πειρατεία τη μοναδική διοκτησία, κλοπή τη διοκτησία. Καθημερινά τα αντιμετωπίζουμε αυτά. Δεν είναι μόνο λοιπόν προστασία του ιδιωτικού βίου, είναι προστασία του μέλλοντό μα, τη δυνατότητα να είμαστε καινοτόμοι στο μέλλον. Εάν δεν προστατεύσουμε τη δυνατότητά μα να ανανεώμαστε στο μέλλον, είμαστε καταδικασμένοι ω κοινότητα. Could you state your name? Hello again. Uh, Το ερώτημά μου απευθύνεται στην κυρία Μάλμστρομ. Αφορά τον εξυγχρονισμό των ε, μηχανισμών εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία πέντε χρόνια τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν πολλή δουλειά για την τροποποίηση του κανονισμού anti-dumping. Έχουμε πλέον δύο κανονισμούς που αφορούν τον εξχρονισμό αυτών των αμυντικών εργαλείων. Πολλοί κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για προστατευτισμό λόγω έλλειψης ορισμού του ε, σοβαρού και ουσιώδους ε, του όρου της σοβαρής και ουσιώδους ε, διαστρέβλωσης του ανταγωνισμού στον κανονισμό. Θέλω και τη δική σας απάντηση. Αν και αν αυτές οι τροποποιήσεις ε, συνάδουν και με, τον, με τους κανόνες του ΠΟΕ. Αυτή είναι η βασική κατηγορία που απευθύνουν χώρες όπως η Κίνα, όπου ήταν, που ήταν η πρώτη χώρα για την οποία συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση. Δεν ξέρω ότι είναι τόσες πολλές ε, οι χώρες που μας κατηγορούν. Η Κίνα σίγουρα, αλλά το, αν υπάρχουν και άλλες δεν το γνωρίζω. Εμείς κάναμε αυτό το εξυγχρονισμό για να ξεκαθαρίσουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιήσουμε, για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, την συμπερίληψη, να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και μάλιστα κατόπιν αιτήματο των κρατών μελών. Ήταν ένας κανονισμός ε, τον οποίο ενέκριναν οι συνομοθέτες. Ξέρουμε ότι η Κίνα μας ε, προσέφυγε εναντίον μα μάλλον στον ΠΟΕ. Θα δούμε πώ θα ε, ποια θα είναι η έκβαση αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρει ποτέ στον ΠΟΕ. Πάντω, εμεί όταν θεσπίζουμε νομοθεσία και όχι μόνο στην εμπορικό τομέα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνάδει και να συμμορφώνεται η νομοθεσία αυτή και με το διεθνέ δίκαιο. Αυτή είναι και η αφετηρία μα. Εμεί θεωρούμε ότι συμμορφώνεται ο κανονισμό μα με το διεθνέ δίκαιο. Εντάξει, κάποια χώρα προσέβηκε εναντίον μα, αλλά πούμε στο δικαστήριο. Αλλά να σα πω την αλήθεια, εμεί έχουμε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση για αυτά που έχουμε κάνει. Ένα ερώτημα που σχετίζεται με αυτό και με την Κίνα, αν δεν κάνω λάθο. Έχετε κι εσεί ερώτηση, Όχι. Ο συντονιστής σχετικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι προσπάθησε να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας, να, διατηρηθούν, ε, να διατηρηθεί ένα ορισμένο επίπεδο επαφών και μέσω τριμερών ε, πρωτοβουλειών που ανέλαβε, προσπάθησε όμως να έχει και διμερείς συζήτηση με την Κίνα. Το ερώτημα μου είναι, πώς μπορεί κανείς να κατακτήσει αυτήν την, αυτόν, αυτήν την μέση οδό ε, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα που έχουν ε, οι σχέσεις ΙΠΑ και Κίνας. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η θέση σας. Πώς, μπορείτε να λειτουργήσετε και ως γέφυρα, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσετε και τις διμερείς σας σχέσεις και με τους δύο εταίρους. Δεν θέλουμε καθόλου να αναγκαστούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στις ΙΠΑ και στην Κίνα, γιατί δεν πρόκειται περί αυτούς, αυτού. Εμείς θέλουμε ένα πολυμερές σύστημα. Για ιστορικούς βεβαίως και οικονομικούς λόγους είμαστε πολύ πιο κοντά με τη ΣΥΠΑ και βεβαίως συμμεριζόμαστε κάποια, κάποια από την κριτική που απευθύνει η ΕΠΑ στην Κίνα. Διαφωνούμε όμως με τις μεθόδους που μετέρχονται. Θεωρούμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το πολυμερές σύστημα. Αν με κάποιον τρόπο λοιπόν μπορούμε να, να μεσολαβήσουμε ώστε οι δύο χώρες αυτές να αρχίσουν ξανά το διάλογο, τότε αυτό ευχή έργων θα ήταν. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο σχέδιο δεν θα έχουμε. Θα ήταν πάντω ευχή έργων, ξαναλέω, να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν τα θέματα για τα οποία διαφωνούν. Όπω είπατε, έχουμε σχέσει και με τι δύο πλευρέ. Ε, είναι διαφορετικέ, βεβαίω, με τον έναν και με τον άλλον. Ωστόσο, βεβαίω και εμεί μπορούμε να προσφύγουμε στον ΠΟΕ όταν θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο, όταν θεωρούμε ότι πλήττονται τα δικαιώματά μα και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε τις επαφές μας και τον διάλογό μας με αυτές τις χώρες στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Βεβαίως δεν έχουμε αυταπάτη ότι εμείς θα είμαστε οι μεγάλοι διαμεσολαβητές που θα λύσουν τα πάντα. Αν όμως έχουμε κάποιες ευκαιρίες στα χέρια μας για να τους φέρουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν, βεβαίω και θα τι αξιοποιήσουμε. Αν και δεν βλέπω αυτό να γίνεται στο άμεσο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας. Κύριε Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά το ποτήρι δεν είναι ακριβώς μισογεμάτο. Πρέπει να συνεχιστεί το έργο και πέρα της κοινοβουλευτικής θητείας, της τρέχουσας, για ακόμη με περισσότερες βελτιώσεις. Μία από τις ιδέες που ε, τονίστηκε πολύ συχνά σήμερα στις τοποθετήσεις είναι η συνέπεια και η συνοχή με άλλους ε, μηχανισμούς και άλλα εργαλεία μέσα που έχουμε δημιουργήσει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, συνοχή και συνέπεια με τους κανόνες μας για τα ανθρωπίνα δικαιώματα με τις αντίστοιχες συμφωνίες που έχουν συναφθεί σε επίπεδο ΟΗΕ, με τους ε, στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ε, για τα εγχώρια μέτρα που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Ταμείο για την Προσαρμογή. Ίσως θα μπορούσε ένας ε, μελλοντικός τίτλος του μηχανισμού που συζητούμε σήμερα να είναι «Εμπόριο για όλους και συνέπεια και συνοχή». Ακριβώς γιατί ε, δεν είναι, το εμπόριο είναι μόνο μία από τις διαστάσεις που μας απασχολούν. Εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ θετική και ενδιαφέρουσα η σημερινή συζήτηση, καθόλου βαρετή νομίζω δεν ήταν. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, φοιτητέ που ήταν σήμερα μαζί μας από τα δύο αυτά πανεπιστήμια. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και για εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές μας και ιδίως βεβαίως τον συντονιστή μας και την επίτροπό μας που ήταν εδώ σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας. Με τα μέλη της Επιτροπής μας θα ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί στις 9. Για όλους του υπόλοιπου, σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο του έτους. Γεια σας.